Se prendete posto possiamo cominciare. Παρακαλώ καθίστε. Σας καλωσορίζω. Μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές έχουμε μια συνεδρίαση για τις επόμενες, ε, τη σημερινή και την αυριανή μέρα οι οποίες είναι θα έλεγα πολύ γεμάτες και γι' αυτό σας προτείνω να υιοθετήσετε την ημερήσια διάταξη έτσι όπως έχει ανακοινωθεί ήδη και αν δεν υπάρχουν διαφωνία σας προτείνω να δεχθείτε τα πρακτικά των συναδριάσεων 4η Ιουνίου, η Ιουνίου, η Ιουλίου και 12 η Ιουλίου. Εντάξει. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Φαίνεται ότι από ε, σε τεχνικό επίπεδο υπάρχουν κάποια προβλήματα με ε, τα πρακτικά, αλλά θα τα διορθώσουμε. Ταυτόχρονα σας θυμίζω ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι αύριο και κλεισμένων των θυρών στις 5.30 θα συνεδριάσουν οι συντονιστές. Υπήρξαν ορισμένα προβλήματα και ο εισαγγελέα Λαουντάτη που έπρεπε να ακούσουμε σήμερα το απόγευμα δεν θα μπορέσει να πάρει το λόγο όπως προεβλέπετο στα πλαίσια του θέματος που αφορά την διαφθορά στον αθλητικό χώρο και θα σας προτείνω κάποιες αλλαγές από τις 5 και 4 μέχρι τις 5.30 θα ακούσουμε τον κύριο Χρυσικό, ο οποίος ε, εκπροσωπεί το UNODC. Και από τις 5.30 ε, μέχρι τις 6 θα ακούσουμε την κυρία Μποσκούρτ, η οποία είναι η εισηγήτρια υπεύθυνη για θέματα αθλητισμού. Εάν συμφωνείτε λοιπόν, έτσι έχει το πρόγραμμα. Ξεκινάμε με το πρώτο σύνολο των συζητήσεων λοιπόν. Είναι η τέταρτη συνεδρίασή μας σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Θα δώσω το λόγο στον καθηγητή κύριο Μιτσιλέγκα, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Eh, Έλεγα λοιπόν ότι είναι μια συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει. Έχετε 15 λεπτά στη διάθεσή σα για να παρουσιάσετε το θέμα σα και μετά θα δώσω το λόγο για δύο λεπτά στου συναδέλφου συντονιστέ και εισηγητέ κυρίω. Αν καταφέρουμε και αν πράγματι καταφέρουμε να σεβαστούμε το πλαίσιο αυτό, μπορεί να υπάρξει και ένας δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Δίνω αμέσως το λόγο λοιπόν στον κύριο καθηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που παρευρίσκομαι εδώ και που θα απευθυνθώ στην Επιτροπή και θα συζητήσω κάποια κύρια ζητήματα σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές παρεμβάσεις στον τομέα του οργανωμένου κλίματος. μου ζήτησαν να συζητήσουμε μια προηγούμενη έκθεση που προετοιμάσα για το Κοινοβούλιο, αξιολόγηση της απόφασης πλαισίου του 2008 και την ποινικοποίηση της συμμετοχής στην κλιματική οργάνωση και να δούμε τι μπορεί να γίνει για να βελτιώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα του οργανωμένου κλίματος. Έτσι λοιπόν, στα 15 λεπτά που έχω σήμερα θα κάνω τέσσερα πράγματα. Καταρχήν, θα συζητήσω μαζί σας το περιεχόμενο, μάλλον το πλαίσιο και την αναγκαιότητα της νομοθέτησης κατά το οργανωμένο κλίματος, κυρίως ε, στον ποινικό τομέα. Το δεύτερο που θέλω να πράξω είναι πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω μια αξιολόγηση για το που βρισκόμαστε σήμερα με την απόφαση πλαίσιο. Το τρίτο είναι να προτείνω κάποια πολύ συγκεκριμένα βήματα. Θα ήθελα να σας ζητήσω να σταματήσετε, λέει η Πρόεδρος. Ε, νόμιζα ότι είναι μόνο το δικό μου ακουστικό, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Στα Ιταλικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την Ιταλική διαρμηνία. Υπάρχει μάλλον, υπάρχουν κάποια παράσιτα, κάποια παρεμβολή. Τώρα, εντάξει. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι μόνο δικό μου το πρόβλημα, αλλά μάλλον προέρχεται το πρόβλημα μόνο από την Ιταλική καμπίνα. Μπορείτε να συνεχίσετε. Με συγχωρείτε. Όπως σας έλεγα, πολύ σύντομα, θέλω να κάνω τέσσερα πράγματα. Καταρχήν είναι να συζητήσω το περιεχόμενο, και την αναγκαιότητα της νομοθέτησης κατά του οργανωμένου κλίματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο είναι να αξιολογήσουμε την απόφαση πλαίσιο του 2008 και να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα, σε ποιο βαθμό ολοκλήρωση βρισκόμαστε στον τομέα αυτό. Το τρίτο που θέλω να συζητήσω μαζί σας είναι το πώς ε, θα προωθήσουμε περαιτέρω την απόφαση πλαίσιο του 2008, τι βήματα μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο. Και το τέταρτο είναι μια ευρύτερη ανάλυση των δυνατοτήτων που προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας για να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο κατά του οργανωμένου κλίματος. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσω να παραμείνω στα 15 λεπτά. Το πρώτο σημείο σε σχέση με το περιεχόμενο και την αναγκαιότητα. Αντιμετωπίζουμε σήμερα ένα παράδοξο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Αφενός, η ανάγκη καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος ε, ήταν η κινητήριος δύναμη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης σε ποινικά θέματα. Κυρίως αν δείτε τη διαδρομή της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης ε, το 1990, θα δείτε ότι πολλά από αυτά που έχουμε τώρα, τον τρίτο πυλώνα, την υιοθέτηση του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και θέτηση νομοθεσία για ευρωπαϊκού οργανισμού στον τομέα αιτιολογήθηκε εν μέρη ε, λόγω τη ανάγκη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. Από την άλλη πλευρά, αυτή η πολιτική όθηση και αυτή η πολιτική ορμή δεν έχει μεταφραστεί σε πάρα πολύ ε, σαφή αναπτυγμένα νομικά πρότυπα κατά του οργανωμένου εγκλήματο. Έχουμε αυτό το παράδοξο λοιπόν αφενό. Υπάρχει μια συνένεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει κάτι για να καταπολεμήσει το οργανωμένο εγκλήματο, αλλά όταν ε, μιλάμε για την ε, μετάφραση αυτού σε συγκεκριμένα μέτρα νομοθετικά, εκεί είναι η πρόκληση. Και τι θέλω να προτείνω στην Επιτροπή. Όταν ε, εξετάζετε πώς θα νομοθετήσετε στο μέλλον πρέπει να συζητηθεί γιατί χρειαζόμαστε νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποιε είναι οι λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου και γιατί θέλουμε να ποινικοποιήσουμε τη συμμετοχή σε μια εγκληματική οργάνωση. Έχω κατηγοροποιήσει αυτές τις λειτουργίες σε πέντε διαφορετικές λειτουργίες της ποινικοποίηση, δηλαδή γιατί θέλουμε να ποινικοποιήσουμε τη συμμετοχή σε μια εγκληματική οργάνωση. Η πρώτη λειτουργία είναι η ανάγκη να ενδυναμώσουμε το εθνικό ποινικό δίκαιο εναντί του οργανωμένου εγκληματός ε, και να έχουν ε, οι εισαγγελείς ένα καλύτερο πλωστάσιο σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα του νόμου, κυρίω ε, στοχεύοντα σε κρατη όπου δεν έχει αναπτυχθεί μια τέτοια νομοθεσία. Αυτό πράγματι θέλουμε να κάνουμε. Είναι ο πρωταρχικός μας στόχο, η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματο. και αυτό σε διαφοροποίηση από άλλα ποινικά δικήματα που μπορεί να εμπίπτουν εκεί. Δηλαδή το οργανωμένο εγκλήμα, έγκλημα προσθέτει κάποια αξία ε, στο να ποινικοποιήσουμε την ε, εμπορία ναρκωτικών ή τη διαφθορά. Ως τέτοιο γιατί θέλουμε να έχουμε ένα αδίκημα πρόσθετο, δηλαδή τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Νομίζω αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να συζητηθεί. Η δεύτερη λειτουργία που μπορεί να εχουμε ενα αδικημα προσθετο δηλαδη τη συμμετοχη σε εγκληματικη οργανωση νομιζω αυτο ειναι ενα ερωτημα που πρεπει να συζητηθει δευτερη λειτουργια που μπορει να εχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στον τομέα είναι να αποσαφηνίσει την εντολή των ε, ευρωπαϊκών οργάνων στην ποινική δικαιοσύνη. Ξέρουμε και η Europol και η Eurojust είναι υπεύθυνοι οργανισμοί για το είναι έρευνα και το συντονισμό της διεθνούς δράσης του οργανωμένου έγκλημα. Αν έχουμε όμως ένα σαφή νομικό ορισμό για το τι σημαίνει το οργανωμένο έγκλημα, τότε προκύπτουν πολλά ερωτηματικά σε σχέση με το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η συνεργασία μεταξύ αυτών των ευρωπαϊκών οργανισμών. Η τρίτη λειτουργία είναι προσπαθούμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι πρόκειται για μια σοβαρή εγκληματική συμπεριφορά η οποία οδηγεί σε αύξηση των ποινών για τα σχετικά εγκλήματα. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε επιβαρυντική περίσταση στο όργανο και τη διάπραξη άλλων αδικηματών. Δηλαδή, χρειάζεται να ποινικοποιήσουμε τη συμμετοχή ε, σε εγκληματική οργάνωση για να τιμωρήσουμε πιο αυστηρά άλλα δικήματα. Τέταρτον, ε, να έχουμε αυστηρές ποινές, ε, αυστηρές κυρώσεις. Μπορεί να είδατε τις πρόσθετες πρόσφατες προτάσεις της Κομισιόν ε, για την κατάσχεση των εσόδων ε, που προέρχονται από το έγκλημα και το οργανωμένο έγκλημα είναι μέσα στην εντολή ε, και έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε το ποινικό δίκαιο για να έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες στον τομέα της κατάσχεσης. Αυτό είναι σημαντικό. Και κάτι άλλο το πέμπτο, που συχνά το έχουμε παραβλέψει, ότι πρέπει να έχουμε σαφήνεια σε σχέση με την ποινικοποίηση του ε, οργανωμένου εγκλήματο ε, για να διευκολύνουμε τη λειτουργία τη αμοιβαία αναγνώριση. Ξέρουμε ότι λειτουργεί πλήρω ε, το ένταλμα το ευρωπαϊκό ένταλμα και επίση έχουμε και την εφαρμογή του νεμπισινίντεμ με e του διτού αξιοπίνου στην Ευρωπαϊκή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως να έχουμε μία ομαλή συνεργασία αν δεν υπάρχει μία κοινή κατανόηση των δικημάτων αυτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα πραγματικό θέμα και βλέπουμε ότι τα εθνικά δικαστήρια συνεχώς αντιμετωπίζουν υποθέσεις όπου κάτι θεωρείται οργανωμένο έγκλημα σε ένα κράτο μέλος αλλά όχι σε κάποιο άλλο. Και οι δικαστές αναρωτιούνται και στέλνουν ε, ερωτήματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να αποσαφηνίσει και αυτό γιατί είναι σαφές το σημερινό πλαίσιο πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η έκτη λειτουργία τέλος που είναι μια ευρύτερη λειτουργία αλλά είναι πολύ σημαντική είναι η θεσμική λειτουργία της ποινικοποίησης του οργανωμένου κλίματος. Η καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος, να χρησιμοποιήσουμε το οργανωμένο κλίμα σε εργαλείο για να διασφαλίσουμε την αμεροληψία, την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος στα κράτη-μέλη. Έχουμε δει σε πρόσφατα κράτη-μέλη ε, προβλήματα στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Κυρίω στη Βουλγαρία την παρακολουθούν ε, για το αν σέβεται τι απαιτήσει κατά πολέμηση του οργανωμένου κλίματο. Πρέπει πέρα από αυτό από την καταπολέμηση, να δυσφανίσουμε ότι έχουμε και εξάρτητο δικαστικό σώμα που μπορεί να εφαρμόσει ε, την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο ποινικό τομέα. Αυτέ είναι οι έξι λειτουργίε. Τώρα που βρισκόμαστε. Η απόφαση πλαίσιο σήμερα έχει αρκετές ελλείψεις και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια δικαίου και το κατά τα θεμελιώδη δικαιώματα και σε ό,τι αφορά στο επίπεδο εναρμόνιση ε, που θα επιθυμούσαμε στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματο, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια δικαίου. Ο τρόπος που έχει διατυπωθεί είναι μια απόπειρα να μεταφραστεί μια ε, προσέγγιση εγκληματολογική μέσα στην νομοθεσία. Τελικά έχουμε πολύ ευρύς ορισμούς για το τι αποτελεί εγκληματική οργάνωση και αν διαβάσετε το άρθρο σχετικά με τον ορισμό της εγκληματικής οργάνωσης στην απόφαση πλαίσιο θα δείτε ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θεωρεί ότι πρόκειται για μια διαρθρωμένη οργάνωση, αλλά αν διαβάσετε την ίδια την παράγραφο θα σας πει ότι δεν χρειάζεται τελικά να είναι και τόσο διαρθρωμένη. Είναι λοιπόν διαρθρωμένη, αλλά δεν χρειάζεται να είναι ιεραρχική. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί σκόπιμα έχουμε έλλειψη σαφήνεια ε, προκειμένου να συμπεριληφθούν πολλέ μορφέ οργανωμένου κλίματο. Αλλά από νομική σκοπιά δεν είναι σε αυτά τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, είμαι σίγουρη ότι η Επιτροπή έχει συζητήσει ότι η απόφαση πλαίσιο ε, προβλέπει και την ποινικοποίηση τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αλλά και την συνωμοσία. Και αυτό είναι το μοντέλο που υιοθετήθηκε επίση από τη Σύμβαση του Παλέρμο για το Διεθνέ οργανωμένο έγκλημα. Η Κομισιόν έχει ήδη αντίρρηση σε αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το εξετάσουμε υπό το φως των διαφορών λειτουργιών της νομοθεσίας ε, που ήδη σας ανέφερα. Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε νομοθεσία στο πλήσιο του οργανωμένου κλίματος. Ποιος είναι ο στόχος ε, να έχουμε αυτές τις ε, δύο εναλλακτικές και Τώρα, σε σχέση με την αξιολόγηση της απόφασης ε, πλαισίου, ξέρω ότι η Κομισιόν ε, στηρίζεται σε διάφορες ε, εκθέσει αξιολόγησης. Τώρα δεν έχουμε βέβαια απαντήσεις. Αλλά θα σα πω τα εξή. Καταρχήν πρέπει να εξετάσουμε πώς τα κράτη-μέλη εφάρμοσαν την απόφαση πλαίσιο, αλλά όχι μόνο σε ό,τι αφορά την νομοθεσία. Δεν αρκεί νομίζω να δούμε το αν υπάρχει ένα νομοθετικό εργαλείο σε κάθε κράτος μέλος που να εφαρμόζει την απόφαση πλαίσιο. Πρέπει να δούμε πώς ε, ε, όσοι εφαρμόζουν το νόμο κατανοούν την έννοια των οργανωμένων κλίματος εισαγγελής, το χρησιμοποίησαν στην πράξη ή όχι. Υπάρχουν ε, σχετικές υποθέσεις δικαστικές για το θέμα αυτό τι έχουν πει τα δικαστήρια για τον οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχει σύγκληση στην ερμηνεία της έννοιας από τα δικαστήρια ή όχι. Οι εισαγγελείς προτιμούν ε, να, να σκούν ε, δίωξη βάσει άλλων ε, αδικημάτων που υπόκειται στο οργανωμένο έγκλημα, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, παραδείγματο χάρη, και αφήνουν κατά μέρο το οργανωμένο έγκλημα. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει μια ποιοτική αξιολόγηση της εφαρμογής της απόφασης πλησίου προκειμένου να αξιολογήσουμε ποια ήταν η προστομένη αξία της απόφασης πλαισίου και αν τροποποιηθεί, προς τα ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να τροποποιηθεί. Η έννοια της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση είναι κατεχρήσιμο ή πρέπει να επικεντρωθούμε σε πιο συγκεκριμένα αδικήματα. Αυτό είναι ένα κεντρικό ερώτημα. Το δεύτερο βήμα προς τα μπρος την άποψή μου και θα καλούσα την Επιτροπή να ζητήσει σχόλια από τα σχετικού οργανισμού. Είναι να υπάρξουν λεπτομερίε ενημερώσει από Europol και για το πώ αυτέ εννοούν την έννοια του οργανωμένου εγκλήματο, αν ο τρόπο που εργάζονται, αν παραδείγματο χάρη αξιολόγηση απειλών από την Europol χρησιμοποιεί τα νομικά κριτήρια που έχουμε στην απόφαση πλαίσιο ή όχι. Ποια είναι η προσταμένη αξία για αυτές τις υπηρεσίες, για αυτούς τους οργανισμούς να έχουν ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία, ποινική νομοθεσία. Είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο, για σε ποιο βαθμό και αυτό είναι σημαντικό. Πώς δηλαδή η Eurojust κατανοεί το οργανωμένο έγκλημα και τι κάνει καθημερινά η Eurojust όταν συντονίζει τους εθνικούς εισαγγελείς για το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος. Ξέρετε, ίσως θα ήταν καλό να διαρνήσουμε περαιτέρω αυτά τα θέματα, δηλαδή τι συμβαίνει στην πράξη επιτόπου. Ένα λεπτό μου έμεινε μόνο για να μιλήσω για τη συνθήκη τη Λισαβόνα, αλλά μπορούμε να τη συζητήσουμε περαιτέρω. Η συνθήκη τη Λισαβόνα δίνει μια σειρά δυνατοτήτων στου νομοθέτε για το οργανωμένο έγκλημα. Καταρχήν, έχουμε το άρθρο 83, παράγραφο 1 τη Συνθήκη Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί συμπεριλαμβάνεται το οργανωμένο έγκλημα και αναφέρεται ρητά ω ένα από το τομεί όπου έχει αρμοδιότητα η Ένωση για να νομοθετήσει. Η ερώτηση νομίζω για την Επιτροπή είναι αν αυτό σημαίνει ότι ε, το, εννοούμε το οργανωμένο έγκλημα αφηρημένο είναι ευστράκτο ή θα πρέπει πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα ποινικά δικήματα όταν έχουν διαπραχθεί στα πλαίσια μιας εγκληματική οργάνωσης. Αυτό νομίζω είναι ένα κύριο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Επίσης έχουμε και το άρθρο 53 παράγραφος 2 και αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο κατά την άποψή μου γιατί εδώ μπορεί να έχουμε ποινικοποίηση τη συμπεριφορά ε, που ε, τελικά μπορεί να ε, ζημιώνει την εφαρμογή άλλων πολιτικών της Ένωσης. Έτσι λοιπόν μπορεί να έχουμε νομοθεσία που να ποινικοποιεί σχετικά δικαιώματα από το οργανωμένο έγκλημα, παραδείγματος χάρη όταν μιλάμε για δημόσιες συμβάσεις. Και ε, τελικά μπορεί αυτό να μην εμπίπτει απευθεία στο οργανωμένο έγκλημα, μπορεί να σχετιστεί με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και ένα άλλο θέμα που θα μπορούσε να διερευνηθεί στο μέλλον είναι η χρήση του άρθρου 86 για τη δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Συγγελικού Γραφείου. Το άρθρο 86 86-4 δίνει δυνατότητα στο μέλλον να ανοίξει εντολή του Συγγελέα για να συμπεριληφθούν και δικημάτα πέρα από την απάτη κατά του προπολογισμού τη Ένωση. Εκεί μπορεί να ε, συμπεριληφθεί και το οργανωμένο έγκλημα. Ξεπέρασε το χρόνο κατά 37 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά που σεβαστήκατε το χρόνο σας και αμέσως θα προχωρήσουμε στη συζήτηση. Ο κάθε παρεμβαίνων θα έχει δύο λεπτά και δίνω το λόγο, θα δώσω το λόγο στη συνέχεια ή στον καθηγητή. Τώρα ο κύριος Νιούτον ε, Τζον. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αντιλαμβάνομαι ότι θα μπορούσατε να μας πείτε ακόμη ε, περισσότερα παρόλο που ξεπεράσατε κατά 30 δευτερόλεπτα και ε, επίσης θεωρώ ότι ε, όντως χρειαζόμαστε κοινοτική νομοθεσία ε, ποινική διότι είναι διασυνοριακά τα ποινικά αυτά αδικήματα οπότε έχουμε εγκλήματα διασυνοριακά τα, κάτι πιο πρόβλημα υπάρχει με τα γαλλικά, παρακαλώ περιμένετε ένα λεπτό γιατί έχουν πρόβλημα με τη διερμηνία στα γαλλικά. Ah, ecco, mi dicono che le tre postazioni della console della cabina Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και στις τρεις θέσεις, στα τρία μικρόφωνα της γαλλικής καμπίνας. Con le, con le cabine, Allora, possiamo vedere se è possibile magari un... Να δούμε... Α, τώρα είμαστε εντάξει. Ωραία. Ξεκινάμε θα παρακαλώ να ξαναξεκινήσετε διότι η, γαλλική καμπίνα δεν μπόρεσε να μεταφράσει αυτά που είπατε. Ευχαριστώ. Ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον καθηγητή. Μπορούσε να μας έχει πει πολύ περισσότερα από ό,τι αντιλαμβάνουμε, από ό,τι του επέτρεπε ο χρόνος του. Θέλω να προτείνω και να τον ρωτήσω αν κατά τη γνώμη του έχω δίκιο ή όχι, ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή νομοθεσία ποινική κατά αυτών των εγκλημάτων είναι ε, διότι ε, ε, είναι όπως το παράδειγμα του, της Μπόνι και Κλάιντ που χρειάστηκε να δημιουργηθεί ομοσπονδιακή νομοθεσία στην Αμερική κατά αυτών των εγκλημάτων διότι ε, άλλαζαν πολιτείες για να διαπράξουν τα δικήματά τους. Το ίδιο λοιπόν ρωτάω πρέπει να γίνει τώρα στον κυβερνοχώρο για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και αν αυτό θα εμπλέξει τη το FBI θα, αν θα εμπλέξει ε, τις φυλακές και πρέπει του χρόνου που θα έχουμε τις συστάσεις να γνωρίζουμε τι θα χρειαστούμε για να βελτιώσουμε την Ευρώπη από αυτή τη σκοπιά και να μας κάνετε τις προτάσεις σας. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Δίας Δεμέρα, για δύο λεπτά για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρους ε, του ΕΛΚ, ε, περιστασίων ε, ελπίζω η Βερονίκα να μπορέσει να το κάνει σύντομα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μητσλεκά που παρευρίσκεται εδώ σήμερα στην Επιτροπή μας. Έχω κάποια σχόλια να κάνω. Εσείς ε, μιλήσατε για έναν ε, πιο αυστηρό ορισμό των εγκληματικών οργανώσεων, δηλαδή να ορίσουμε καλύτερα τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση. Όμως εγώ θα ήθελα να σας πω ότι από πρακτική σκοπιά ο ορισμός αυτός ε, δεν έχει και ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, δεν έχει πολλά αποτελέσματα και μάλιστα είναι αδύνατο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά να εναρμονίσουμε τους ποινικού κώδικες γιατί έχουμε διαφορετικούς νομικούς πολιτισμούς, έχουμε ρίζες λατινικές και ρίζες εκλοσαξονικές σε κάποια κρατημέλη όπως γνωρίζετε και σε κάτι που είναι πτέσμα σε ένα κράτος μέλος, σε ένα άλλο κράτος μέλος μπορεί να είναι πλημέλημα. Έτσι λοιπόν είναι δύσκολο να οδηγηθούμε βρεθούμε στο δρόμο αυτής της εναρμόνισης. Και τώρα σε σχέση με την Ευρωπόλ, όπως ξέρετε, έχει μία νομική βάση που βασίζεται σε μία απόφαση του Συμβουλίου. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκόλμης και το πρόγραμμα των δράσης, ε, είναι ότι σε λίγες μέρες αυτό το κοινοβούλιο θα ασχοληθεί, θα συζητήσει τον κανονισμό που θα καλύψει νομικά τη Europol. Εσείς νομίζετε, πιστεύετε ότι μπορούμε σε αυτό το νέο κανονισμό να αντιμετωπίσουμε την περιπέτεια να παράξουμε έναν πιο αυστηρό ορισμό για τις εγκληματικές οργανώσεις και τέλος, ε, να σας πω ότι είμαι απόλυτα σκεπτικός σε όσα λέγονται στα άρθρα 84 και 86 της Συνθήκης της Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την αναφορά σε ένα σε ένα γραφείο εισαγγελικό. Γιατί είμαι σκεπτισκιστής, γιατί το Συμβούλιο συστηματικά κάθε φορά που το Κοινοβούλιο κάνει λόγο για κάτι τέτοιο, το Συμβούλιο στρίβει το κεφάλι από την άλλη. Αυτά και σας ευχαριστώ. Θα να μου σχολιάσετε τόσο σας ανέφερα. Ε, ε, ευχαριστώ. Τώρα, φαγιό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο καθηγητή για τις εξηγήσεις που έδωσε. Σίγουρα θα μπορούσατε να μας πείτε πολύ περισσότερα. Βέβαια βιώνουμε όπως είπατε ένα παράδοξο σήμερα. Από τη μία όλοι θα συμφωνήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει περισσότερα στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος. Απ' την άλλη όμως οι κυβερνήσεις θα πρέπει επιτέλους να αναλάβουν δράσεις απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις. Είναι σαφές ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι απειλή για την ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία. Ιδιαίτερα στα πλαίσια της κρίσης, της οικονομικής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει βρει νέα εδάφη, ιδιαίτερα για τις συμμορίες της οργανωμένες όπως η μαφία. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει μια πιο συνολική αντιμετώπιση και στον τομέα της πρόληψης και στον τομέα της επιβολής του νόμου. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό ορισμό του οργανωμένου εγκλήματος. Εφόσον το πετύχουμε κάτι τέτοιο θα βοηθήσει, θα συνεισφέρει στην πρόληψη του οργανωμένου εγκλήματος και σε επίπεδο διαμεθοριακό. Το θέμα είναι να δούμε πόσο βλέπει κανείς την υπάρχουσα μορφή λειτουργία του Europol και της Eurojust. Έχετε μια γενική άποψη για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι υπηρεσίες αυτές θα έχουμε και ακροάσεις με εκπροσώπους αυτών των οργανώσεων και έτσι ίσως μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την άποψή μας για το πώς φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους. Πώς αντιμετωπίζετε την κριτική που ασκείται από τις κυβερνήσεις για τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών. Έχουν λόγο ύπαρξης, φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε και ένα Ευρωπαίο εισαγγελέα. Αναφερθήκατε σε αυτό, αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Κομισιόν στην ομιλία του στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα λοιπόν και τη δική σας άποψη, πώς βλέπετε τα πράγματα στον τομέα σας. Η πολιτική μας ομάδα, στην πολιτική μας ομάδα, τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, εμένουμε ε, στο να γίνει μια σωστή μελέτη του αν πράγματι έχει νόημα η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Ευχαρίστως έχω γράψει και σημείωσα τα άρθρα τα οποία θεωρείτε ότι είναι χρήσιμα από την Λισαβόνα 3.1, 83.2 και νομίζω ότι είπατε ότι υπάρχει κι άλλο ένα άρθρο που μπορεί να επιτρέψει την ε, ένταξη, δηλαδή το 64. Θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε ότι σας μιλώ για το σωστό άρθρο. Όσον αφορά τα κράτη-μέλη, νομίζω ότι υπάρχει ήδη υποδομή. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές νομοθεσίες ε, ε, όσον αφορά το ποινικό δίκαιο ε, στα διάφορα κράτη-μέλη και εδώ διαφοροποιούμε από τον Ισπανό συνάδελφο, αλλά όλοι νομίζω αντιμετωπίζουμε τη διαφθορά με τον ίδιο τρόπο. Πήγαμε και στη Σερβία και θεωρούμε ότι η διαφθορά είναι εξίσου σοβαρό αδίκημα ε, παντού σε όλες τις χώρες και ακόμη και αν δεν ε, υπάρχει οργανωμένο έγκλημα υπάρχει διαφθορά και η διαφθορά είναι ε, ένας τομέας που θέλουμε να πατάξουμε. Γι' αυτό και νομίζω ότι καλό θα ήταν να γίνει αυτό το οποίο είπατε, δηλαδή να υπάρξει περισσότερη και καλύτερη ποιοτική αξιολόγηση. Ίσως σήμερα αργότερα ή αύριο μπορεί να μας ε, γίνει ε, ε, κάποια ενημέρωση σχετικά με την ποιοτική αξιολόγηση. Δηλαδή να ξεχωρίσουμε τι δεν είναι άμεσα διασυνοριακή εγκληματικότητα αλλά από πλευράς νομικής κατανόησης και αποθελήσεως πατάξεως ιδίως για τα νέα κράτη που προσχωρούν όπως κάποια μέρα η Σερβία και η Κροατία θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή αυτή η ποιοτική αξιολόγηση την οποία ζήτησε ο καθηγητής θα ήθελα να ξέρω αν μπορεί στην Επιτροπή μας να δοθεί και να θεωρηθεί σαν μια έμπειρη γνώμη. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση πριν δώσω το λόγο στον ε, καθηγητή όσο είπε ο κύριος Δίας μέρα προηγουμένως είναι αληθή ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε έναν ε, ενιαίο ορισμό για το οργανωμένο έγκλημα. Όχι μόνο γιατί πρέπει να περάσουμε από την αρμόνιση όλων ε, των νομικών συστημάτων, κάτι που ήδη είναι αρκετά δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και ε, ελληπής πολιτική βούληση. Γιατί ε, αυτό γίνεται αντιληπτό μόνο σε συγκεκριμένε χρονικέ στιγμές. Όλοι θα θυμόμαστε ότι μία από τι πρώτε προτεραιότητε που τέθηκαν στην έκθεση που εθετήσαμε τον Οκτώβριο του 2008, δηλαδή την έκθεση με τον οργανωμένο έγκλημα, μία από τι προτεραιότητε ήταν να θεωρηθεί η απόφαση του Συμβουλίου του 2008, η απόφαση πλαίσιο, γιατί υπάρχει ο κίνδυνο, ε, μια ε, ερμηνεία αφηρημένη και τελικά να μην λέει τίποτα η συνάδελφος Φαγιών είπε ότι το οργανωμένο έγκλημα απειλεί την οικονομία των χωρών μας. Εγώ θα πρόσθετο ότι απειλεί και την ελευθερία και την ασφάλεια 550 εκατομμυρίων πολιτών. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια δέσμευση. Uh, uh, uh, τα κράτη-μέλη πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι πέρα από τα λόγια. Αυτή είναι μια πτυχή που μπορούμε να την αγγίξουμε πρακτικά κάθε φορά που έχουμε σοβαρά επιχειρηματά. Υπάρχουν μεγάλα προγράμματα, όλοι συμφωνούμε, αλλά κατόπιν ε, όταν ε, θα ε, πρέπει να ε, κάνουμε κάτι στην πράξη, στο κοινοβούλιο, αρχίζουν να δυσκολεύουν τα πράγματα. Θέλω, θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε εσείς για το ρόλο της Ευρωπόλ και βάσει και της αναθεώρησης της νομικής βάσης. Εσείς δεν θεωρείτε ότι είναι σκόπιμο τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν να επενδύσουν πραγματικά στο ρόλο της Ευρωπόλ και να θεωρηθεί η Ευρωπόλ ως μια δομή που θα μπορούσε να έχει ουσιαστικά ένα ε, ρόλο ανταλλαγής πληροφοριών, παραδείγματο χάρη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες που προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά υπάρχουν και χώρες που το κάνουν εντελώς ε, εικονικά και κατόπιν. Είναι δύσκολο να υπάρξει καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος διασυνοριακά. Εγώ να υπενθυμίσω μόνο το εξή. Ε, είμαι σίγουροι ότι είναι φαινικό, αλλά θέλω να θυμάστε, αν το οργανωμένο έγκλημα έγινε σήμερα η απειλή νούμερο ένα σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι επειδή το οργανωμένο έγκλημα δεν έχει γεωγραφικά σύνορα, δεν έχει νομικέ βάσει να εναρμονίσει. Το οργανωμένο έγκλημα ξέρει πολύ καλά πώ να εναρμονιστεί σε διεθνέ επίπεδο και πώς να ριζώσει στις διάφορες χώρες. Είχαμε και την κυρία Μπορσελίνο που ήθελε το λόγο. Παρακαλώ για δύο λεπτά. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μία παρατήρηση. Έχω την αίσθηση ότι ξεκινήσαμε να μπαίνουμε στην ουσία της συζήτησης για το οργανωμένο έγκλημα γιατί θεωρούμε ότι αυτή η μορφή εγκλήματος είναι υπεύθυνη για μια εν μέρη τουλάχιστον για τη χειροτέρευση της οικονομικής κρίσης στον κόσμο τα συμφέροντα του οργανωμένου εγκλήματος υπονομεύουν ε, μια αγορά η οποία ήδη έχει τα δικά της προβλήματα και την υπονομεύουν και μέσω της ε, στρεβλής, του στρεβλού ανταγωνισμού που ε, κατά κάποιο τρόπο ανταγωνίζεται αυτή η φαιά μορφή της οικονομίας την κανονική αγορά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον μας εκεί. Ίσως θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα να το κάνουμε αυτό, γιατί έχουμε μέσα στη διάθεσή μας. Έχουμε όμως την εντύπωση ότι τα ονόματα, οι τίτλοι Eurojust, Europol στην ουσία είναι κάποιοι πυρήνες απομεμακρυσμένοι και ασυντόνιστοι μεταξύ τους κάνουν τη δουλειά τους αλλά δεν είχαν ουσιαστικό στόχο να αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο συγκεκριμένες καταστάσεις παρανομίας και εγκληματικότητας. Σήμερα μιλάμε για το οργανωμένο έγκλημα αλλά πολλές φορές ακούω στις ομιλίες ότι υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα στην εγκληματικότητα, στη μαφία κτλ. Δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός αυτής της δραστηριότητας, αυτής της κατάστασης. Εγώ νομίζω ότι αν πράγματι θέλουμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό με πραγματικό στόχο το να αντιπαρατεθούμε με το έγκλημα αυτό, απαιτείται ένας ορισμός κοινός ξεκάθαρος για όλους. Παρ' όλα αυτά, αυτή η προσπάθεια εναρμόνισης των διαφόρων ενιών της εγκληματικότητας που εκφράζονται με μια κάποια σύγχυση σήμερα θα πρέπει να περιγράψουν ουσιαστικά μια παράνομη πράξη. Γιατί αν δεν υπάρξει μια τέτοια συγκεκριμένη αναφορά στη δράση των εγκληματικών αυτών δικτύων της μαφίας δεν μπορούμε να επιτεθούμε σε αυτά τα σύνολα ούτε σε ποινικό επίπεδο αλλά ούτε και σε επίπεδο πολιτισμικό θα έλεγα Ήδη έχουμε σε ένα πρώτο επίπεδο μια κάποια μορφή σύγχυσης μπροστά μας και δεν ξέρουμε γιατί, γιατί μιλάμε. Αν κάθε χώρα όμως μιλάει με μια κοινή γλώσσα, αλλά έστω και με τη δική της κλίδα ανάγνωσης, τότε θα έχουμε κάνει κάτι θετικό. Ας ξεκινήσουμε από εκεί λοιπόν και τότε θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις τις οποίες έχουμε μπροστά μας, εφόσον πράγματι έχουμε τη βούληση να αντιπαρατεθούμε με το οργανωμένο έγκλημα με, με, όλες τις μορφές που έχει σαν μια σαφέστατα παράνομη ε, ενέργεια. Ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Το εξετίμησα πάρα πολύ και θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω τις απαντήσεις μου σε τρία βασικά θέματα τα οποία ε, παρουσιάστηκαν από τις ερωτήσεις. Το πρώτο, το οποίο διεφάνει από όλες τις ερωτήσεις οι οποίες ετέθησαν, είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε τον ρόλο των ε, ε, ευρωπαϊκών ε, θεσμικών οργάνων στον ρόλο της καπατάξεως της εγκληματικότητα, ο ρόλος δηλαδή της Europol, της Eurojust, το γραφείο του Ευρωπαίου Ισαγγελέα και ούτω καθεξής. Και Τώρα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη της Λισαβόνας ανοίγει την πόρτα σε μια επανεξέταση του ρόλου αυτών των οργανισμών οι οποίοι ανέπτυξαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανεπτύχθησαν χωρίς κάποια συστηματική ε, διάταξη και βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές επικαλύψεις μεταξύ των εντολών τους και κάποιος ανταγωνισμός μεταξύ των οργανισμών. Τώρα με την συνθήκη της Λισαβόνας όπως είπατε έχουμε μία νέα νομική βάση και πρέπει να δούμε ποιο είναι το όραμά μας. Πώς πώς θέλουμε να, υποκαταστήσουμε ε, τα εθνικά όργανα και πόσο θέλουμε να βοηθήσουμε. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος της Όλαφ παραδείγματος χάρη σε αυτό το σύνολο. Έχει νόημα, αν υπάρχει ένας ε, εισαγγελέας θα πρέπει να συγχωνευτεί με το γραφείο του εισαγγελέα, το ίδιο και με το Eurojust. Τώρα, σχετικά με την Europol, αυτό που είπε η πρόεδρος είναι ότι είναι τόσο καλός οργανισμός όσο η πληροφόρηση που δίδεται από τα κράτη-μέλη. Αλλά αν αποστασιοποιηθούμε πρέπει να δούμε τι θέλουν ε, τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πράττει η, ε, Ευρωπα... Europol. Θέλουμε να είναι συλλογή πληροφοριών ε, για την εγκληματικότητα ή τι. Πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτούμε και να αναρωτηθούμε γιατί έχουμε αυτούς τους οργανισμούς τους ευρωπαϊκούς και τι θέλουμε να κάνουν. Είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει και να δούμε και σε ποιον είναι υπόλογοι ε, ε, όλοι αυτοί οι οργανισμοί. Εξετάζονται πλήρως ποιο είναι το μέλλον των ατόμων που ε, επηρεάζονται από την ύπαρξη αυτών των οργανισμών. Έχουμε παραδείγματο χάρη μία ενδιαφέρουσα περίπτωση με το Λουξεμβούργο και τη δράση της Όλαφ. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι ε, μπορούν να αποτελήσουν βάση για μία έκθεση. Ε, είναι ίσως ε, πιο βασικό να δούμε τι θα κάνουν οι οργανισμοί, βασικότερο και από την νομοθεσία σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα. Όσον αφορά την οργάνωση και την εναρμόνιση. Η εναρμόνιση δεν, εννοεί, δεν υπονοεί ομοιογένεια σε όλα τα κρατη με θέλει Εναρμόνιση, η συνθήκη μιλά για οδηγίες, η οδηγία είναι δεσμευτική ως προς τους στόχους και αφήνει τη διακριτική ευχέρεια στο κράτος να κινηθεί και αυτό είναι πολύ βασικό αλλά για να απαντήσω στα θέματα σχετικά με τον στόχο νομίζω ότι στην απόφαση πλαίσιο έχουμε ένα τόσο ευρύ και ασαφή ορισμό που όχι μόνο ε, θέτει σε κίνδυνο την ε, νομική βεβαιότητα και ασφάλεια αλλά είναι τόσο ευρύς ορισμός ώστε να μην έχει πλέον νόημα. Οπότε πρέπει να σκεφτείτε γιατί θέλετε την νομοθεσία και πώς θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε και να καταλήξετε σε συγκεκριμένους ορισμούς σχετικά με τα θέματα που θέλετε να προωθήσετε. Και το τελευταίο θέμα το οποίο ίσως χάθηκε στην μετάφραση εγώ αναφερόμουν ε, στο άρθρο 86 ε, παράγραφος 4 για τον Ισαγγελέα ε, που ρυθμίζει δηλαδή την την ε, ίδρυση του γραφείου του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και πιστεύω ότι πρέπει να δούμε πόσο οι οργανισμοί και η απόφαση πλαίσιο λειτουργήσαν. Πώς δηλαδή ε, αντιμετώπισαν οι εθνικές αρχές όλα αυτά τα θέματα και συγχρόνως να κάνουμε ε, μία αξιολόγηση για την, ε, τις εθνικές πράξεις και την αξιολόγηση της Europol και της Eurojust. Είναι κάτι που η Επιτροπή σας ίσως θα έπρεπε να ε, επιληφθεί. Δηλαδή δεν αναφερόμαστε μόνο στα κράτη-μέλη και ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν θεματοφύλακα των συνθηκών, αλλά πιστεύω ότι και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ βασικός. Ευχαριστώ τον κύριο καθηγητή. Κλείσαμε λοιπόν το πρώτο σύνολο των συζητήσεων. Θα ξεκινήσουμε με τον δεύτερο κύκλο κυβερνοέγκλημα σαν μέσο της εγκληματικής δραστηριότητας. Θα ακούσουμε μια γαλίδα δικαστή, την κυρία Μυριάμ Κεμενέρ, η οποία είναι εμπειρογνώμων στα θέματα του κυβερνοεγκλήματος. Θα ακούσουμε τον κύριο Σέρλινγκ, εκπρόσωπο της Europol και τον κύριο Χάιμανς από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων. Θα κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνουμε πάντα, 15 λεπτά παρουσίασης μετά θα υπάρξουν δύο λεπτά για τους συντονιστές και μετά θα κάνουν ερωτήσεις οι υπόλοιποι βουλευτές. Δίνω το λόγο αμέσως στην κυρία Κεμενέα για να μας παρουσιάσει την έκθεσή της. Ευχαριστώ Πρόεδρε που με προσκαλέσατε για να αναφερθώ στο κυβέρνο έγκλημα. Μέσα από αυτά τα οποία ήδη ακούστηκαν υπάρχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία ανάμεσα στην οργανωμένη εγκληματικότητα και το κυβερνοέγκλημα. Αναφερθήκαμε στην απουσία ορισμού. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση του ε, κυβερνοεγκλήματος. Τα κείμενα, οι βασικοί νόμοι δεν διευκρινίζουν τα πράγματα ακριβώς. Ένα παράδειγμα, η σύμβαση της ε, Βουδαπέστης αναφέρεται στην εγκληματικότητα στον κυβέρνοχώρο. Τι θα πει κυβέρνοχώρος, είναι κάτι το πάρα πολύ φλού. Είναι λοιπόν μία από τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας για το φαινόμενο και στη Γαλλία και στις υπόλοιπες χώρες, πώς να ορίσουμε ακριβώς το θέμα αυτό. Έχοντας πάρει μέρος σε προσπάθειες εργασίες και στα πλαίσια του GNDC, διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα κανείς τα πράγματα σωστά. Στη Γαλλία έχουμε, δίνουμε μια ευρεία ερμηνεία, μιλάμε για παράνομες δραστηριότητες σε επίπεδο πληροφορικής ή κυβερνοπειρατεία, αλλά ταυτόχρονα και κάποιες ε, παραδοσιακές παράνομες πράξεις όπως οι απάτες, οι, οι ε, προσπάθειες υφαρπαγής ταυτοτήτων που ε, τελούνται μέσω του ψηφιακού μέσου και ταυτόχρονα υπάρχει μια τρίτη κατηγορία αν θέλετε είναι ε, συκοφαντία, ρατσισμός, ε, παιδοφιλία μέσω του διαδικτύου. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχουμε μια κάποια δυσκολία σε σχέση με τον ορισμό της εγκληματικότητας των κυβερνοχώρων. Και αυτό έχει συνέπειες. Στους βασικούς νόμους το θέμα του κυβερνοεγκλήματος δεν ξεκαθαρίζεται στα πλαίσια σαν παράδειγμα του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Αν γίνεται αναφορά βέβαια χωρίς όμως να ορίζεται. Αυτό είναι ένα εμπόδιο και ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να πούμε ότι η δικαιοσύνη μερικές φορές αντιμετωπίζει δυσκολίες στα πλαίσια της διαχείρισης αυτών των των δραστηριοτήτων ε, για μια δραστηριότητα η οποία κατ' εμέ βέβαια είναι μια ε, δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος. Καταρχάς υπάρχει, υπάρχει το θέμα της εξωτερικής δικαιοδοσίας, δηλαδή μια επίθεση κυβερνητική σε μια πολύ μακρινή χώρα μπορεί να έχει επιπτώσεις και στο γαλλικό έδαφος ή στο ευρωπαϊκό έδαφος γενικότερα. Οπότε ποιος είναι ο νόμος που θα εφαρμοστεί εδώ. Υπάρχουν θέματα εδαφικής δικαιοδοσίας. Και υπάρχουν και πάρα πολλά τεχνικά θέματα. Για τους δικαστές απαιτείται ε, ανεξαρτήτως χώρας η οποία εμπλέκεται απαιτούνται συγκεκριμένες μορφές κατάρτισης και στη παρούσα φάση στη Γαλλία γίνονται προσπάθειες κατάρτισης έτσι ώστε οι δικαστές οι οποίοι είναι νομικοί βέβαια να μάθουν τα βασικά της λειτουργίας αυτών των δραστηριοτήτων που επιτρέπουν να τελούνται ενέργειες που συνδέονται με το κυβερνοέγκλημα. Ποιες είναι λοιπόν οι νομικές απαντήσεις. Πώς μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτού του είδους τις παραβατικές δραστηριότητες. Καταρχάς, ο νομοθέτης ε, λαμβάνει υπόψη του την συγκεκριμένη διάσταση δημιουργώντας συγκεκριμένες παράνομες πράξεις σαν παράδειγμα παρεμβάσεις ανεπίτρεπτες στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, παρακράτηση προσωπικών στοιχείων, σύγκληση ε, και δημιουργία ομάδας με εγκληματική δράση και σκοπούς και επίσης ε, έχουν χρησιμοποιηθεί και κάποιες μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί σαν επιβαρυντικά στοιχεία για να κατασταλούν τα φαινόμενα τα σχετικά με την, με την εγκληματικότητα σαν παράδειγμα η παράνομη χρήση ενός δικτύου τηλεπικοινωνιών που επιβαρύνει την επιβολή της ποινή. Γενικά αυτές είναι οι τάσεις. Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να αναφερθούμε στα διαδικαστικά που χρησιμοποιούν τα δικαστήρια με πολύ συγκεκριμένες κάθε φορά δράσεις. Καταρχάς, ο έλεγχος ε, των ε, στοιχείων που προέρχονται από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή από το διαδίκτυο. Υπάρχουν επίσης κάποιες ανακριτικές τεχνικές οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στην ανάγκη καταπολέμησης της ε, εγκληματικότητας σαν παράδειγμα ο εισοδισμός σε εισαγωγικά σε ψηφιακό επίπεδο η χρήση ψευδονύμων για να έρθει κανείς σε επαφή με κάποιον ο οποίος ε, κατηγορείται ή είναι ύποπτος για τέτοιου είδους δράσεις. Άλλες μορφές ανάκρισης και έρευνας οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στον ψηφιακό κόσμο είναι η παρακράτηση δεδομένων από απόσταση, δηλαδή ένας δηλαδη ένα υπευθυνο της εισαγγελία, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα Trojan ένα ένα δούριο ύπο για να μπορέσει να πάρει στοιχεία που θα οδηγήσουν στην διατύπωση μιας κατηγορίας. Η νομοθεσία λοιπόν σε επίπεδο υλικού δικαίου και σε επίπεδο διαδικαστικού δικαίου έχει ήδη προσαρμοστεί αρκετά. Έχουν δημιουργηθεί νέες παράνομες πράξεις όχι μόνο στην Γαλλία αλλά και σε πάρα πολλές άλλες χώρες όπως ε, η υποκλοπή της ταυτότητας online, κάτι το οποίο δημιουργεί ε, στη δημιουργία νέων προφίλ για συμμετοχή με εγκληματικό στόχο στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό που φαίνεται μέσω της προσπάθειας επεξεργασίας αυτής είναι ένα δίκαιο του διαδικτύου με ένα νομικό καθεστώς το οποίο έχει καθοριστεί σε σχέση με τους παροχείς, τους τεχνικούς. Δηλαδή με ελαφρυντικά εκεί υπάρχουν ε, οι, ε, οι ευθύνε τους και εμπλέκονται μόνο από τη στιγμή κατά την οποία τους γνωστοποιούνται κάποιες παράνομες πράξεις που έχουν ήδη τελεστεί μέσω των δικτύων τους. Πρόκειται για ένα καθεστώς ευνοϊκό θα έλεγα για τους παροχείς στα πλαίσια του νόμου για την ψηφιακή οικονομία έτσι ώστε να επιτροπεί η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου αποφεύγοντας όμως τρευλώσεις και καθιστώντας το ασφαλές. Αυτά τα συστήματα λοιπόν ε, ευθύνης με ελαφρυντικά θα έλεγα των παροχέων ε, υφίσταται αρκετή κριτική στη Γαλλία και μερικές φορές γίνονται ορισμένες προτάσεις μέσω σαν παράδειγμα κοινοβουλευτικών προσχεδίων κάποιες προτάσεις για νέα καθεστώτα που αφορούν σαν παράδειγμα αυτό που ονομάζουμε online εκδότης. Δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχουν προτάσεις και για σωστή και ευρυθμι... Ε, λειτουργία των πληστηριασμών εξαποστάσεων. Εξαποστάσεως. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών λοιπόν οι νέοι εταίροι του ε, ίντερνετ του διαδικτύου που έχουν έρθει στην επιφάνεια δεν καλύπτονται πλήρως νομικά. Το ίδιο γίνεται με τα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα σε επίπεδο νομικό. Στην παρούσα φάση στη Γαλλία θεωρούνται σαν απλή, ε, απλή χώρη φιλοξενίας με μειωμένη ευθύνη. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα. Σε επίπεδο δικαστικό, τι άλλο μπορούμε να διαπιστώσουμε, ότι όλο και περισσότερο υπάρχουν πολλές μορφές απάτης οι οποίες γίνονται μέσω των ψηφιακών δικτύων. Πρόκειται για αρκετά περίπλοκες απάτες οι οποίες απαιτούν πολύ συχνά διεθνή συνεργασία. Πρέπει να γίνονται έρευνες και στο εξωτερικό. Ε, υπάρχουν διεθνή εντάλματα ανακριτικά και ε, πολλοί εμπειρογνώμονες έχουμε προτείνει εδώ την χρήση απλούστερων γενικά διαδικαστικών μέσων εκτός από τα συγκεκριμένα αυτά ανακριτικά εντάλματα γιατί το να προσπαθήσουμε να κάνουμε ε, μια σωστή προσπάθεια ε, έρευνας μιας παράνομης δραστηριότητας είναι στην ουσία ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο. Απαιτείται άμεση αντίδραση λοιπόν όταν υποπτευόμεθα μια εγκληματική δράση που προγραμματίζεται να γίνει στο διαδίκτυο. Πολλές φορές τα αιτήματα για τη δημιουργία αυτού του εντάλματος αργούν ε, και απαιτείται χρόνος. Απαιτείται εναρμόνιση λοιπόν και των μέσων συλλογής αποδείξεων Πολλές φορές τα δεδομένα παρακρατούνται στη Γαλλία για ένα χρόνο, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση δύο χρόνια. Υπάρχουν δυσκολίες συντονισμού εδώ και μία από τις δυσκολίες καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος είναι η δυσκολία συλλογής αποδείξεων. Σαν παράδειγμα στις Ηνωμένε Πολιτείες είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ιστοσελίδες για ε, να χρησιμοποιηθούν σαν παγίδα για τους παρανόμους. Στην Γαλλία απαγορεύεται αυτό με τα απόφαση του Αριοπάγου ε, λέγοντας ότι οι αποδείξεις θα πρέπει να συλλέγονται με νόμιμο τρόπο και όχι μέσω στρατηγημάτων και παγίδες ε, δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται. Ε, υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν λοιπόν για την εναρμόνιση της συλλογή των αποδείξεων. Αυτό είναι βασικό. Θα πρέπει επίσης να απλοποιηθούν τα διαδικαστικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να καταλήγουν σωστά οι δικαστικές διαδικασίες γιατί διαπιστώνουμε σήμερα ότι όσο υπάρχει από τη μία μια ενίσχυση των μέσων για τους ανακριτές το βλέπουμε αυτό μέσω ειδικών υπηρεσιών Υπάρχουν ε, ειδικοί ερευνητές αστυνομικοί που ασχολούνται με τα εγκλήματα στον τομέα του διαδικτύου. Αλλά σε επίπεδο δικαστών δεν υπάρχει μια τέτοια ειδίκευση, μόνο σε επίπεδο δικαστικής αστυνομίας. Και πολλά θέματα κυβερνοεγκλήματος γίνονται αντικείμενο αντιμετώπισης από υπηρεσίες που ασχολούνται γενικότερα για το, με το οικονομικό έγκλημα. Βλέπουμε όμως ότι εδώ υπάρχουν δυσκολίες γιατί έχουμε να κάνουμε με διαφορετικούς εμπλεκομένους και εταίρους. Εδώ απαιτείται συνεργασία επίσης και με τον ιδιωτικό τομέα. Σε πάρα πολλές ε, περιπτώσεις χρειάστηκε να συνεργαστούμε με τις νομικές υπηρεσίες πολλών μεγάλων οικονομικών εταιριών οικονομικά μεγάλων ενώ εταιριών και αυτά είναι καινούργιοι τρόποι θα έλεγα λειτουργίας και είναι κάτι με το οποίο δεν είναι πολύ συνηθισμένοι να δουλεύουν τουλάχιστον οι Γάλλοι δικαστές. Κλείνοντας λοιπόν την παρουσίασή μου θα ήθελα να πω ότι ένα από τα βασικά εμπόδια της καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος είναι η έλλειψη ορισμών. Το κυβερνοέγκλημα συνδέεται βέβαια με μια μορφή οργανωμένου εγκλήματος, από την άλλη πρόκειται για κάτι το πάρα πολύ συγκεκριμένο. Είναι κάτι στο οποίο εμπλέκονται συμμετέχοντες και τεχνικοί παροχής οι οποίοι συνεργάζονται όλο και περισσότερο με τους δικαστές. Αυτοί οι παροχείς έχουν σαν παράδειγμα δημιουργήσει υπηρεσίες δικαστικής συνεργασίας για να δίδουν απαντήσεις τάχιστα στα αιτήματα των δικαστηρίων. Το σύστημα αυτό βελτιώνεται και η δικαιοσύνη πολύ όμως εξαρτάται από την καλή βούληση και την γρήγορη ανταπόκριση αυτών των εταίρων. Απαιτείται λοιπόν καλύτερη εναρμόνιση. Απαιτείται επίσης περαιτέρω προσπάθεια κατάρτισης όλων των εμπλεκομένων δικαστών, δικαστική αστυνομία κτλ. και σε επίπεδο πανεπιστημιακό και σε επίπεδο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια, ιδιαίτερα σε τομείς όπως το Ευρωπόλ, το Interpol, το Eurojust. Σχηματικά τα λέω όλα αυτά ότι στα πλαίσια της προσπάθειας ε, της καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος υπάρχει μια διάχυση και σε επίπεδο νομικών βάσεων και σε επίπεδο δομών υπηρεσιών, ανεξάρτητες υπηρεσίες που διαπιστώνουν κάποιες παράνομες δραστηριότητες και τις καταγγέλουν στην εισαγγελία. Αναφέρομαι σαν παράδειγμα στην αρχή εποπτείας των online στοιχημάτων που ε, παραπέμπει κάποιες υποθέσεις στην ε, εισαγγελία στο Παρίσι. Αυτή η αρχή σαν παράδειγμα δεν είναι πάρα πολύ γνωστή σε πολλούς δικαστές και αυτό είναι κάτι το οποίο παρεμποδίζει την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κυβερνο, του κυβερνοεγκλήματος. Υπάρχει επίσης και το ότι σε επίπεδο δικαιοδοσιών ε, έχουν υπάρξει προβλήματα. Εμείς έχουμε προσπαθήσει στα πλαίσια της περιφέρειας του Παρισιού να εργαστούμε με τα δύο βασικά δικαστήρια τα οποία πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους στα πλαίσια ορισμένων χρηστών πρακτικών. Να υπάρχουν κάποιοι θα έλεγα συγκεκριμένοι δικαστές στους οποίους να αναφέρονται και οι εμπλεκόμενοι όλοι και στον τομέα των επιχειρήσεων και στον τομέα των ε, ε, ιδιωτών. Βέβαια αυτές δεν είναι μόνιμες υπηρεσίες, είναι υπηρεσίες ad hoc οι οποίες εξαρτώνται πολύ από τον δυναμισμό των συγκεκριμένων δικαστών. Πρέπει λοιπόν ε, ότι όπως και στις, προηγούμενες, περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι ειδικέ δικαστικές υπηρεσίες θα πρέπει να οργανώνονται σωστά σε κεντρικό επίπεδο. Στη Γαλλία δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σαν παράδειγμα ένας δικαστικός πόλος ψηφιακός στα πλαίσια του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα επέτρεπε να δοθεί μια νέα όθηση και να δημιουργηθεί θα έλεγα μια ουσιαστική ποινική ε, ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων σε επίπεδο ποινικό. Γιατί ένας τέτοιο δικαστικός πόλος θα δίνει συμβουλέ στους δικαστές που έχουν ανάγκη από σωστέ πληροφορίες και ενημέρωση και έτσι θα καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά αυτή τη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος το οποίο είναι κάτι το πάρα πολύ περίπλοκο για τους απλούς δικαστές. Σας ευχαριστούμε για τις εξηγήσεις που μας δώσετε κυρία Κέμερερ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο για 15 λεπτά στον κύριο Τρέλ Σέρτινγκ που εκπροσωπεί την Ευρωπόλη. Παρακαλώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που καλέσατε τη Γεωρόπολη σε αυτή την πολύ σημαντική ακρόαση. Εγώ θα προσπαθήσω να διατηρήσω τη συζήτηση όπως την υλοποιούμε εμείς στην αστυνομία και να σας δώσω κάποιες συμβουλές ε, σε σχέση με το πώς θα έπρεπε να είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Κατεπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του στον κυβερνοχώρο.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 Αν δείτε εδώ τις εξελίξεις, ε, το 1950 υπολογίζαμε το 60 ερευνούσαμε, τη δεκαετία του 70 αρχίσαμε να συνδεόμαστε ένας με τον άλλο και τη δεκαετία του 80 συνεχίσαμε με την επικοινωνία. Τη δεκαετία του 90 αρχίσαμε τη δημοσίευση και τη δεκαετία του 2000 ε, είχαμε το Twitter, το Facebook, το Skype ε, και άλλες υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2010 έχουμε το υπολογιστικό νέφος ε, και δεν ξέρω τι να προβλέψω για το 2020. Και δεν θέλω να προβλέψω τίποτα γιατί τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα θα δείτε στατιστικά στοιχεία. Βλέπετε, εκεί είχαμε 1,8 δισεκατομμύρια το ίντερνετ, 1 δισεκατομμύριο χρήστες του Facebook, Google, ε, πάνω από 1 δισεκατομμύριο καθημερινά επισκέπτες σελίδες μέσω Google, πάνω από 274 δισεκατομμύρια email, καθημερινά στέλνονται και πάνω από 200 δισεκατομμύρια από αυτά είναι spam, ανεπιθύμητα email. Καθημερινά βλέπουμε ε, πάνω από 140 ε, ε, δίκτυα να δημιουργούνται και κάθε δευτερόλεπτο βλέπετε 46 νέους κακόβουλους κώδικες και αυτό είναι το συλλογικό απολογισμός για το κυβερνοέγκλημα. Αλλά μπορώ να εκτιμήσω το οτιδήποτε αν δούμε τώρα το ιστορικό και δούμε τι έγινε ε, το 70 δεν ε, υπάρχει κανένας λόγος ε, κάποιος να θέλει να κάνει προβλέψεις στο σπαμ θα είναι σε δύο χρόνια κάτι που θα ανήκει στο παρελθόν, είπε ο Bill Gates το 2004 και το iPhone δεν έχει κανένα σημαντική, καμία σημαντική ε, δυνατότητα να λάβει μερίδιο στην αγορά αν είχαν πει. Όμως εγώ πώς να προβλέψω το μέλλον όταν, όταν αυτοί οι κύριοι που ήταν εμπειρογνώμενες δεν μπορούσαν να το κάνουν. Τι κρύβεται ε, τελικά πίσω από την ανάπτυξη και την ευημερία στο διαδίκτυο. Αντιμετωπίζουμε μία σειρά προκλήσεων στο μέλλον. Σήμερα ε, έχουμε την εκδοχή 4 του IP, του πρωτοκοποκόλου και σύντομα θα πάμε στην εκδοχή νούμερο 6. Ποια είναι η διαφορά. Σήμερα έχουμε 3,4 δισεκατομμύρια δυνατότητες διευθύνσεων IP, ε, ενώ στην εκδοχή 6 θα έχουμε 2,4 δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια διευθύνσεις. Και η αστυνομία πρέπει να βρει σε ποιον ανήκουν οι διευθύνσεις αυτές. 73% των χρηστών του ίντερνετ δεν χρησιμοποιούν τα αγγλικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι στο 72% ε, των συνδεδεμένων χρησιμοποιούσαμε, έχουμε τα τελευταία πέντε έτη που χρησιμοποιούμε το δίκτυο είχαμε πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ότι τα προηγούμενα 50 χρόνια της βιομηχανικής επανάσταση. Έχουμε ένα τρισεκατομμύριο ε, συσκευών που πωλείται και οι κινητές συσκευές ήδη το περισσότερο από τα PC, από τους υπολογιστές. Αν ε, πάρετε ε, τώρα την παλιά μπαταρία του δικού μου Mac και τη βάλετε στο καινούριο, δύο λεπτά θα κρατήσει. Αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη των δυνάμεων των μπαταριών και των, και των ισχύω ε, των κομπιούτερ Σε αυτή την περιοχή του κόσμου που έχουμε δυσκολίε και έχουμε λιτότητα, δεν είμαστε μια τεράστια βιομηχανική περιοχή, δεν παράγουμε με τον παλιωμοδίτικο τρόπο πλέον αγαθά, ήδη τα αγαθά παράγονται σε περιοχές όπου κοστίζει αυτό να Όμω Εμεί εφευρίσκουμε, έχουμε έρευνα και ανάπτυξη, έχουμε διαχείριση της ε, αλυσίδας εφοδιασμού, μπορεί κάποιος να κατεβάσει βιβλία από τι ε, ηλεκτρονικέ βιβλιοθήκε αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα αναπτυχθούμε και θα έχουμε την ευμερία αν το επιτρέψουμε και να το φροντίσουμε. Αλλά επίσης υπάρχουν και νέοι κίνδυνοι και ο κυβερνοχώρος ε, πάντοτε το έκανε αυτό και θα το εκμεταλλευτούν τρομοκράτες, ακτιβιστές, εγκληματικές ομάδες αλλά και μυστικές υπηρεσίες ξένες και δεν ε, υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι μύθος. Δεν μπορούμε να ασφαλίσουμε τα πάντα στο διαδίκτυο αν έχετε ένα πάρα πολύ σημαντικό έγγραφο με τη συνταγή της Coca-Cola, μην το βάλετε στο ίντερνετ γιατί θα το βρουν. Αλλά φυσικά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από ό,τι κάνουμε σήμερα. Οι διοκτικές αρχές αντιμετωπίζουν νομικές προκλήσεις σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα. Η Γαλλίδα συνάδελφος μόλις μας ενημέρωσε ότι πρέπει να επιταχύνουμε αυτή τη δουλειά και συμφωνώ απόλυτα. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα αργότερα. Τώρα, ποιε είναι οι προκλήσει. Ε, καταρχήν, πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιου κανόνε αλλά και ευαισθητοποίηση αν μπορούμε να χρησιμοποιήσω ένα καθημερινό παράδειγμα, αν είναι κάποιος ε, πολύ μεθυσμένος ε, και ε, κάνετε βόλτα στο κέντρο του Άμστερνταμ, στο με το πορτοφόλι σας ανοιχτό, μάλλον θα σας κλέψουν. Και το ίδιο είναι αν κάνει κάποιος περιπελία σε μέρη που δεν πρέπει να πάει, ή μάλλον συγγνώμη, αν κάποιος μπαίνει σε κακές ιστοσελίδε, τότε κάποιοι θα επιτεθούν στον υπολογιστή του. Έτσι λοιπόν ότι είναι παράνομο στον πραγματικό κόσμο θα πρέπει να είναι παράνομο και στον επιγραμμικό κόσμο και ε, πρέπει τώρα να προστατεύσουμε 550 εκατομμύρια ανθρώπους σε 27 κράτη-μέλη με 23 διαφορετικές γλώσσες και επίσης διαφορετικά νομικά συστήματα και πρέπει να επικεντρωθούμε στο οργανωμένο έγκλημα γιατί υπάρχει μια τάση κάποιοι όλοι χάρη ε, να θέλουν να προωθήσουν όλε τι ψηφιακέ ε, κλοπέ στο διαδίκτυο τον των ποδηλάτων λόγου χάρη δεν χρειάζεται να επικεντρωνόμαστε στα πάντα παραδείγματο χάρη. Μια άλλη απειλή που βλέπουμε τώρα ε, στη Europol είναι τέσσερις μεγάλοι τομεί. Καταρχήν εισβολή, ε, δεύτερον απάτη, κατόπιν ε, ε, έχουμε την κλοπή προσωπικών δεδομένων και επίσης την εκμετάλλευση των παιδιών και αυτό δυστυχώς αυξάνεται. θα αναφερθώ σε μια χώρα, δεν θα αναφέρω το όνομά της, αλλά αυτή η χώρα είχε δύο χρόνια καθυστέρηση ε, για ε, καταγγελίες ε, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και είχε πει ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι λοιπόν η ψηφιακή παραοικονομία. Όλα στο διαδίκτυο σημαίνουν χρήμα θα μπορούσε να είναι πληροφορίες για ταυτότητά σας, οι πιστοτικές σας κάρτες, άλλοι τομείς και θα μπορούσαν όλα αυτά να δημιουργήσουν, να παράξουν χρήμα. Εμείς αυτό αξιολογούμε το επιχειρηματικό μοντέλο του ε, εγκλήματος στον χώρο. Αν ε, το δείτε, είναι κάτι που λειτουργεί από πάνω προς τα κάτω. Μια υπάρχουν κάποιοι κωδικοί ε, και υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται για να κλέβουν τους κωδικούς, κατόπιν υπάρχουν άλλοι πιο κάτω και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που ουσιαστικά εκτελούν, κλέβουν αυτά που θέλουν να κλέψουν. Τότε δεσμεύει το οργανωμένο για να κλέψει τα χρήματά σου, αγοράζει κάτι κάτι και στη συνέχεια αφαιρεί τα χρήματα. Δείτε αυτή την αλυσίδα ε, του επιχειρηματικού μοντέλου και συγκρίνεται το με την κανονική δουλειά που κάνει η αστυνομία. Αν είχαμε παραδείγματο χάρη ε, στοιχεία να καταπολεμήσουμε το κοκαίνι, ξέρετε ότι παράγεται κοκαίνι στην Νότια Αμερική, κατόπιν πρέπει ε, να συλλεχθεί, θα πρέπει να πάει στα δικαστήρια, να κοπεί, να μπλεχθεί με πρόδρομέ ουσίε και πρέπει να πάει στην Κολομβία, να σταλεί συνήθω στην Ισπανία Γερμανία και από την Ισπανία συνήθως ε, μοιράζεται σε μικρές μερίδε ε, και εδώ θα τη βρείτε στη συνέχεια στην πλατεία, στι Βρυξέλλε ή στο Παρίσι. Δείτε αυτή τη μεγάλη γραμμή όπου η αστυνομία έχει πάρα πολλές πολλε δυνατοτητε να δράσει. Όμως ε, αυτό το έγκλημα μπορεί να γίνει σε ένα υπόγειο με έναν υπολογιστή. Δεν υπάρχουν ίχνη, ούτε υπάρχουν σύνορα να περάσει κανεί, ούτε υπάρχουν ευάλωτα σημεία. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσει η αστυνομία. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντριο Καταπολέμησης των Κλίματος στον ε, κυβερνοχώρο ε, θέλει να ασχοληθεί και με τους χάκερα, αλλά και με όσου ξεπλένουν ε, τα χρήματα. Η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο δεν θα είναι ένα τμήμα αυτών των τομέων γιατί το κυβερνοέγκλημα είναι, για τον κυβερνόμενο είναι πολύ δύσκολο να δούμε ποιο είναι το κίνητρο. Αν δούμε μία επίθεση στον κυβερνοχώρο, μπορεί παραδείγματο χάρη να είναι από πίσω ένας 16χρονος ακτιβιστής, μπορεί να είναι ε, κάποιος που ανήκει σε τρομοκρατική οργάνωση ή σε οργάνωση οργανωμένου κλίματος. Αυτό δεν μπορούμε να το δούμε. Ε, και Γι' αυτό θα πρέπει όλες ε, οι κατασταλτικές υπηρεσίες να εργάζονται μαζί, γιατί πρέπει να κατανοούμε που δραστηριοποιείται ο καθένα, Η Κομισιόν θέλει εμείς στη Europol μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013, πολύ σύντομα δηλαδή, να ιδρύσουμε ένα ευρωπαϊκό κέντρο κατά πολεμή των κλίματο στον κυβέρνοχώρο. Η Europol επιλέχθη για αυτή τη δουλειά γιατί έχουμε ένα εύρωστο σύστημα που ήδη λειτουργεί και αυτό θέλουμε να παράξουμε ως αποτέλεσμα και έχω το προνόμιο να είμαι ο πρώτος επικεφαλής ε, του κέντρου. Θα αναλάβω τα καθήκοντά μου την 1η Ιανουαρίου και ελπίζουμε να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες ε, στις αστυνομικές υπηρεσίες στα κράτη-μέλη. Καταρχήν, να έχουμε ένα κέντρο παροχής πληροφοριών, δηλαδή να ενημερώνει για το τι συμβαίνει εκεί, γιατί το έγκλημα στον κυβερνοχώρο δεν συνδέεται με ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό τόπο, δεν είναι ότι έγινε μια ληστεία εδώ ή ένα βιασμό μπορεί να έχει γίνει, σε ένα υπόγειο στη Γερμανία, το θύμα να είναι στη Σουηδία και να έχει χρησιμοποιηθεί ένα σερβερ στην Ινδία. Πρέπει να έχουμε μια επισκόπηση για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη για να μην κάνουν διπλή προσπάθεια σε κάθε περίπτωση. Θα δημιουργήσουμε και ένα ε, κέντρο για να βοηθήσουμε τις ε, αστυνομικέ αρχέ των κρατών μελών να εργαστούν μαζί σε μια κοινή ερευνητική ομάδα. Θα προσφέρουμε και επιχειρησιακή υποστήριξη, κάτι που ήδη συμβαίνει σε διάφορες υποθέσεις και εγκληματολογική υποστήριξη. Πρέπει να σας πω ότι σε πάρα πολλά από τα κράτη-μέλη, κυρίως τα μικρότερα κράτη-μέλη, δεν υπάρχει ο προπολογισμό για τέτοια εγκληματολογικά εργαλεία. Δεν υπάρχει. Και αντί να δημιουργηθεί ένα σύστημα σε 27 κράτη-μέλη ε, για να βρουν το ίδιο εργαλείο και 27, το δικό μας το κέντρο θα πάρει όλε αυτέ τι απαιτήσει και ελπίζουμε να πείσουμε την Κομισιόν να δώσει κάποια κονδύλια για να αναπτύξουμε αυτά τα εργαλεία και να τα δώσουμε στα κράτη-μέλη. Ελπίζω ε, θα καταρτήσουμε του αστυνομικού, του εισαγγελεί και του δικαστέ και ένας από τους ε, τομείς αυτών των δυνατοτήτων είναι να προσθέσουμε τις ε, ζωτικές υποδομές στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και επίσης να υπάρχει και σύμπραξη ιδιωτικού δημοσίου τομέα και θα πρέπει να έχουμε και έκθεση σοβαρών περιστατικών και να τις εξετάσουμε. Και τέλος, σε ποιον ανήκει το ίντερνετ, σε κανέναν δεν ανήκει το ίντερνετ. Ποιος ρυθμίζει το διαδίκτυο. Κυρίως δύο φορείς, το ICAN και η ITU. Ε, η ICAN ε, είναι ένας εταίρος ιδιώτης στον οποίο ανήκουν όλα τα δικαιώματα για τις ονομασίες και για τις διευθύνσεις IP και ETU. είναι μια οντότητα των Ηνωμένων Εθνών που εργάζεται σε αυτό το τομέα. Αλλά για τις διοκτικές αρχές είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε εμεί μια φωνή έτσι ώστε αν βλέπουμε να διαπράτεται το έγκλημα και υπάρχει η δυνατότητα ε, να μπορέσουμε να βρούμε τους δράστες διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτό το κέντρο ε, είμαστε ε, ιδιαίτερα συμπεριληπτικοί. Ακούσαμε ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των διαφορών υπηρεσιών, διαφορών οργανισμών. Δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός ε, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για το έγκλημα στον χώρο. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει τόσο πολύ έγκλημα που αρκεί για όλους. Έτσι λοιπόν τι χρειάζεται να κάνουμε. Απλώς να συντονίσουμε τις προσπαθίες μας ε, και να δημιουργήσουμε συνέργειες, ε, να... Ε, βασιστούμε σε όσους κάνουν ήδη μια εξαιρετική δουλειά. Έτσι λοιπόν ήδη ε, η Eurojust θα έχει ένα γραφείο σε εμάς, η Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης κτλ. Δεν θα υπάρχουν επικαλύψεις αλλά καλύτερη επισκόπηση και επίσης θα έχουμε και εταίρους σημαντικούς Τώρα, ε, στη Σιγκαπούρη υλοποιείται ένα ψηφιακό κέντρο που θα είναι έτοιμο το 2015 και θα επικεντρωθούν στο παγκόσμιο κυβερνοεγκλήμα. Θα ανταγωνιστούμε. Όχι, εγώ κάλεσα τον κύριο Σανακατάνη, ο οποίο είναι επικεφαλή αυτή τη οντότητα, να συμμετέχει και στο δικό μα συμβούλιο και θα υπάρχει πλήρη διαφάνεια. Θα ξέρει τι θα κάνει η Europol ε, και μαζί με ε, τη δική του οντότητα θα συνεργαστούμε για να έχουμε ένα παγκόσμιο αντίκτυπο και θα λειτουργήσουμε από κοινού. Η οικονομία είναι κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μύθο ότι είναι ε, δυνατό να καταπληρώσουμε το κυβερνό έγκλημα. Είναι δύσκολο, δεν είναι αδύνατο και ε, δεν έχουμε προσπαθήσει ακόμα στην πραγματικότητα. Φυσικά δεν θα είναι δωρεάν, αλλά αξίζει να επενδύσουμε σε αυτό. Σεβάστηκα το χρόνο μου και μάλιστα έκανα και πέντε δευτερόλεπτα λιγότερο. Σα ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ κύριε Όρτινγκ. Θα δώσω το λόγο τώρα για 15 λεπτά στον κύριο Χάιμανς, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι που μας καλέσατε και μετά τη Europol είδαμε πόσο, πόσα εγκλήματα υπάρχουν να καταπολεμηθούν και πόσο βασική είναι η συνεργασία όπως είπε ο κύριος Σούτεγκ ε, και αυτό περιλαμβάνει και τις αρχές ε, προστασίας των δεδομένων και αυτή θα είναι η δικιά μου συμβολή και ίσως για όσους δεν γνωρίζουν τη θέση του επόπτη για την προστασία ε, δεδομένων ε, είμαστε ε, ο οργανισμός που εποπτεύει όλες τις νέες νομοθεσίες και εγώ από τη θέση μου Προσφάτως σχολίασα το Ευρωπαϊκό Κέντρο για ε, εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Γιατί είναι τόσο βασική η προστασία των δεδομένων και γιατί είναι ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Διότι η καταπολέμηση του ε, εγκλήματος στον κυβερνοχώρο ε, συνεπάγεται προστασία προσωπικών δεδομένων και εισδοχή στον ιδιωτικό χώρο των πολιτών διότι για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα στον κυβερνοχώρο ε, πρέπει παραστατικά να ε, προσπαθήσουμε να συνδέσουμε το έγκλημα με άτομα και ενδεχομένως με άτομα τα οποία μέχρι τώρα δεν ε, θεωρούνται καθόλου ύποπτα για εγκλήματα μία αποτελεσματική στρατηγική για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος που ε, θέλω να παρουσιάσω δεν μπορεί ε, να υπάρξει χωρίς να συνοδεύεται από μια γερή προστασία των ε, δεδομένων θέλω να αναφερθώ και στο σύστημα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται από τις διοκτικές αρχές και από τους εποπτικούς οργανισμούς για το διαδίκτυο όπου παρακολουθούν και ε, διώκουν ε, τις εγκληματικές πράξεις. Είναι βέβαια χρήσιμο να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες ε, για προστασία δεδομένων. Έχουμε διάφορους ορισμούς που υπέβαλαν ε, προλαλήσαντες ε, ομιλητές και που είναι αποτελεσματικές αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ξέρουμε περισσότερο τι είναι το κυβερνοέγκλημα διότι για μας υπάρχουν ουσιαστικά δύο διαφορετικά εγκλήματα τα οποία προσπαθούμε να διαφοροποιήσουμε. Καταρχήν ε, ε, τα δικήματα ε, κατά του διαδικτύου των υπολογιστών η κλοπή, η παραχάραξη οτιδήποτε δηλαδή μειώνει την ασφάλεια ενός συστήματος ε, και επίσης από την άλλη πλευρά υπάρχει το παράνομο περιεχόμενο διότι το περιεχόμενο αυτό ε, είναι καταρχήν ε, εγκληματικό και επίσης υπάρχει και παράνομη αποδοχή στοιχείων από το διαδίκτυο downloading οπότε ε, πολλές φορές η πράξη είναι αυτή η οποία ε, ε, πλήττει την προστασία των δεδομένων εάν υπάρχει ένας hacker από το facebook από κοινωνικά μέσα ενημέρωσης ή από τραπεζικούς λογαριασμούς από πλευράς προστασίας του των δεδομένων ε, ο τομέας αυτός είναι πάρα πολύ προβληματικός διότι για να καταπολεμήσουμε το ε, ε, κυβερνοέγκλημα πολλές φορές χρειαζόμαστε τη βοήθεια και τη συνδρομή των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών και αυτοί εμπλέκονται στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και πρέπει να κάνουν πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το βασικό τους καθήκον να διαθέτουν πληροφορίες και να υπάρχει ε, ουδετερότης, δηλαδή να μην επεμβαίνουν οι υπάροχοι. Ε, στην περίπτωση όμως αυτή πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο. Μιλάμε για την παρακολούθηση του διαδικτύου. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται για να είμαστε αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και τελευταίος έχουμε ε, συμμετάσχει και σε διαδικασίες όπου η παροχή ενημερώνονται ότι υπάρχει παράνομο κατέβασμα πληροφοριών ε, με προστατευμένη πνευματική διοκτησία και πρέπει να κλείσουν ορισμένες ιστοσελίδες. Αυτή λοιπόν ε, η, ε, αυτό το θέμα είναι απαραίτητο για την προστασία των δεδομένων και επηρεάζει την ουσία της προστασίας δεδομένων, δηλαδή να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά μόνο για τον αρχικό στόχο τους και όχι για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος. Όλα αυτά βέβαια είναι περιορισμένα, δεν είναι απεριόριστα και ελεύθερα. Όταν όμως μιλάτε για εμπλοκή των υπευθύνων των διαδικτύων και ε, των διοκτικών αρχών ε, ε, είναι βασικό να υπάρχει μία αναλογικότητα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να υπάρξουν, εάν ε, μιλάμε ε, παραδείγματος χάρη νόμος ε, για θέματα όπως η παιδική πονογραφία πρέπει να προστατεύσουμε και τα δικαιώματα των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων και εδώ η αναλογικότητα είναι πολύ σημαντική σχετικά με την εφαρμόσιμη νομοθεσία για προστασία δεδομένων όπως σας είπα υπάρχει μία νομοθεσία η οποία έχει κατοχυρωθεί στο άρθρο 8 του χάρτη των βασικών δικαιωμάτων όπου λέγεται ότι όλοι έχουν δικαίωμα να προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Όλα τα στοιχεία αυτά πρέπει να τα χειρίζεται κανείς ε, με ε, συγκεκριμένο τρόπο και ο καθένας έχει έχει δικαίωμα να ξέρει τι είναι, ποια είναι η τύχη των δεδομένων που έχουν συλλεγεί γύρω του και η διαφάνεια είναι επίσης βασική για την προστασία των δεδομένων κατά τρόπον ώστε να ελέγχουμε τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα. Αυτά δεν είναι τόσο δύσκολα. Μετά όμως ερχόμαστε στο θέμα του πού εφαρμόζει την νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και εδώ αντιμετωπίζουμε προβλήματα ε, όταν μιλάμε για κυβερνοέγκλημα διότι οι δικαστικές ε, ε, και αστυνομικές αρχές καλύπτονται στον τρίτο πυλώνα και η καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος είναι ένα θέμα που δεν είναι εύκολο να οριοθετηθεί. Υπάρχει μια γενική απόφαση πλαίσιο του 2008 υπαριθμών 997 και υπάρχουν και συγκεκριμένοι κανόνες. Είναι όμως δύσκολο να γνωρίζουμε ποιο ποιος είναι ακριβώς ο κανόνας, ο που εφαρμόζεται. Η Europol έχει το δικό της σύστημα και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ε, ε, αυτού. Όταν φτάνετε ε, στον ρόλο των ISPs, των ε, ε, παρόχων ε, διαδικτυακών υπηρεσιών τότε τα δεν ξέρουμε αν καλύπτονται από τα άρθρα του πρώτου πληλώνα 95-46 ή από κάποιο άλλο σημείο. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει δυσχεράνει την κατάσταση και δεν έχει διευκολύνει να διευκρινιστεί. Τώρα λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται στο Συμβούλιο και εδώ νομίζω ότι ο εισηγητής παρακολουθεί. Ελπίζω ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια Ιδίω για τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών όταν είναι υποχρεωμένοι να συνδράμουν τις διοκτικές αρχές αλλά παραμένουν δεσμευμένοι από τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Τώρα θα ήθελα να πω ότι η προστασία των δεδομένων και είναι κάτι που έχω επαναλάβει πολλές φορές η προστασία δεδομένων βοηθά να εντοπίσουμε κινδύνους και ε, προβλέπει όταν ε, καταρτίζεται ένα σύστημα στο κτίριο της Europol για τον κυβερνοχώρο η ιδιωτική πτυχή πρέπει να ληφθεί υπόψη από την αρχή και θα πρέπει να είμαστε, είμαστε υπόλογοι όταν αναπτύσσουμε μία τέτοια προστασία δεδομένων εξού και έχουμε συνεργαστεί σε ένα πρότυπο ανταλλαγής στοιχείων για να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα στοιχεία έχουν ληφθεί υπόψη οι χρήστες. Πρέπει επίσης να εξοδοτηθούν. Η προστασία αυτή είναι επίσης σημαντική και πέραν αυτού οι οργανώσεις πρέπει να εξασφαλίσουν τις γέφυρας προστασίες δεδομένων που να επιτρέψουν να είναι αποτελεσματική η καταπολέμηση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Και τώρα έχουμε στην συνεργασία των παρόχων ε, διαδικτυακών υπηρεσιών με τις διοκτικές αρχές. Χρειάζεται πολλές φορές η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα διότι ε, ε, αυτοί έχουν τα στοιχεία, όχι η αστυνομία και αυτό είναι περίπλοκο διότι ουσιαστικά αυτό το οποίο μας ανησυχεί από αυτή την οπτική γωνία είναι ότι δεν πρέπει να φτάσουμε σε ένα σύστημα όπου συστηματικά ε, όλοι πρέπει να παρακολουθούν συστηματικά ό,τι γίνεται στο διαδίκτυο διότι η συστηματική παρακολούθηση του διαδικτύου είναι πολύ επεμβατική ενώ υπάρχουν και νομικές υποχρεώσεις ή απαγορεύσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο παραδείγματος χάρη όπου υπάρχουν υποχρεώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών αλλά υπάρχει η ε, οδηγία 2258 η οποία απαγορεύει τη συστηματική παρακολούθηση του, ε, του, του δικτύου από τους παρόχους. Βάσει του, της σάκτα βάσει της ε, ουδετερότητος και της αναγνωρίσεως ε, του χαρακτήρα των ε, δεδομένων αυτών προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση για να παρακολουθούμε το κυβερνοέγκλημα που έχει μεγάλη έκταση όπως είπε ο προλαλής σας. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται ε, είναι ε, να υπάρχει μία γενική παρακολούθηση των πληροφοριών που διακινούνται και το δικαστήριο είπε ότι θα πρέπει κανείς ε, να συμβιβάσει τα διάφορα συμφέροντα και δεν πρέπει να είμαστε επεμβατικοί και να μπαίνουμε σε θέματα που δεν έχουν άμεση σχέση με το θέμα μας. Νομίζω ότι στα κέντρα πατάξεως του κυβερνοεγκλήματος χρειάζεται να υπάρχει αυτή η προστασία και στις συστάσεις μας προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε ορισμένα σημεία πιστεύουμε όμως γενικότερα ότι η πρόληψη είναι ένα θέμα ε, όπου ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε και να προβλέπεται την προστασία των δεδομένων εις ε, την ε, καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος. Έχω ελάχιστο χρόνο για τα συμπεράσματά μας. Όπως σας είπα, πρέπει να αποφύγουμε τη συστηματική παρακολούθηση. Ε, ο συστηματικός εντοπισμός των χρηστών είναι μία σαφής παραβίαση των ε, βασικών νομικών αρχών. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε συστηματική παρακολούθηση του περιεχομένου του διαδικτύου. Ε, νέα κέντρα θα πρέπει από την αρχή να εφαρμόζουν τους κανόνες προστασίας των δεδομένων. Θα πρέπει η προστασία να είναι αντίστοιχη με το στόχο μας και γι' αυτό ζήτησα από τις ε, ε, διοκτικές και τις δικαστικές αρχές να είναι πολύ προσεκτικές για να μην παραβιάζουν τα βασικά δικαιώματα των ατόμων. Ευχαριστώ κύριε Χάιμανς. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Ο κύριος Διέστε Μέρα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτό το πλήρες και πολύ ενδιαφέρον πάνελ. Ευχαριστώ τους τρεις ε, ομιλητές, ε, την κυρία Κεμενέρ, τον κύριο Χίσμαν ε, και τον κύριο Έκτη, για τη συνεισφορά τους. Δεν θα κάνω ερωτήσεις, απλώς θα κάνω μια ερμηνεία της πραγματικότητας και του προβλήματος που έχουμε ενώπιόν μας, που είναι πώς να καταπολεμήσουμε ε, τα αντικείμενα που σχετίζονται με το γνωμένο έγκλημα. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να βρούμε μια νομική ισορροπία μεταξύ της ερευνητικής διαδικασίας και της προστασίας ε, της ιδιωτικής ζωής. Δηλαδή πρέπει να πετύχουμε πάντα αυτή την ε, νομική ισορροπία. Και εγώ νομίζω ότι για να καταπολεμήσουμε την κλοπή ταυτότητας, την ε, απάτη, την παιδεραστία και την τρομοκρατία υπάρχει μια σειρά στοιχείων που τίθεται εδώ επιτάπητος και των οποίων η ερμηνεία δεν ε, είναι εύκολη αυτά με ένα συνοπτικό τρόπο το παρουσιάζω καθώς ε, πιο γρήγορα προχωρά το έγκλημα από τη δικαιοσύνη αλλά στο κυβερνοέγκλημα αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο, η ταχύτητα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Αυτά είναι πολύπλοκα θέματα αλλά εγώ θα τα απλοποιήσω. Για το αδίκημα ή ε, δικαστές είπαν ότι χρειάζονται ειδικές δομές. Εσείς είστε ειδικοί, αλλά πόσους ε, ειδικούς δικαστές ε, έχετε στην Γαλλία ένα δεύτερο στοιχείο, μία ταχεία δράση ε, και πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Εμείς οι νομοθέτες είμαστε πάρα πολύ αργοί και οι εγκληματίες είναι πολύ γρήγοροι. Κατόπιν έχουμε το θέμα και του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου. Αυτό είναι πολύπλοκο θέμα, ιδιαίτερα πολύπλοκο, γιατί δεν ε, υπάρχει ε, ε, δεν σέβονται την νομοθεσία με πάρα πολλές προφάσεις και πολλές φορές ε, οι προφάσεις αυτές έχουν οικονομική θεμελίωση. Αυτά είναι γνωστά. Δεν ε, χρειάζεται να δώσω εγώ τώρα στοιχεία που όλοι μπορεί να γνωρίζουν. Όμως, από την άλλη πλευρά, καθώς υπόκειται και στην νομοθεσία, στον νόμο, μπορεί να επικαλεστούν την οδηγία προστασία των δεδομένων όποτε του χρειάζεται. Αυτό είναι ένα νομικό κενό ιδιαίτερα πολύπλοκο. Βέβαια, η προστασία των δεδομένων παρέχει εγγύσεις αλλά επίσης και η καταπολέμηση του εγκλήματος, δηλαδή οι διοκτικές αρχές χρησιμοποιούν παρανομικά εργαλεία για να υπάρξει αστυνομική δίσδυση. Και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Είναι ένα θέμα που δεν έχει επιληθεί και δεν το λέω εγώ έτσι χωρίς να μου κοστίζει. Και τέλος, υπάρχει ένα θέμα που δεν θίξαμε εδώ, αλλά υπάρχει στον αέρα και υπάρχει στο ε, κυβερνοχώρο που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ξέρετε, ε, μιλάμε για ε, τις ε, παρακολουθήσεις, ε, παραδείγματος χάρη μπορεί να υπάρχουν κάποιοι πομποί που να μπουν στο αυτοκίνητο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι μπορεί κάποιος να ακούσει και να αποκτήσει ιδιωτικές πληροφορίες. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα, ιδιαίτερα ισχυρά και οι δημοκρατίες ακόμη δεν είμαστε σε θέση να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, να τις εξοδετερώσουμε. Γι' αυτό με ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό το τελευταίο θέμα που θίξατε, που έχει να κάνει με τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα ε, των διοκτικών αρχών. Ε, και τώρα θα έχουμε και συνεργασία ε, και Χάγης. Να δούμε πώς θα τα ε, οργανώσουμε όλα αυτά. Πρέπει να ολοκληρώσει τηλεπρόεδρος. Ναι, ναι, ναι, ολοκλήρωσα. Μίλησα ήδη πολύ καιρό. Νομίζω ότι αρκούν τα όσα είπα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. σα. ευχαριστώ για την υπομονή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τους φιλελεύθερους, ο κύριος Νιούτον Ντάν. Ευχαριστώ και τους τρεις ε, ομιλητές. Ε, πράγματι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις, αν και υποχρεωτικά ενοχλητικά σύντομες. Να πω σωστά τα ονόματά σας. Για την κυρία Κεμενέρ καταρχάς. Μας είπατε ότι η παγίδευση είναι παράνομη στην Γαλλία. Εγώ ε, συναντήθηκα με έναν Βέλγο αστυνομικό ο οποίος μου είπε το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και να έλθω τώρα στην παρουσίαση του κ. Χάιμαντς. Εσείς θα υποστηρίξετε μια αλλαγή του νόμου για την παγίδευση στο διαδίκτυο, να είναι εφικτή η παγίδευση για την αστυνομία. Γιατί κάτι τέτοιο απαγορεύεται λόγω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εγκληματιών. Βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες το FBI μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, φρικτά πράγματα εις βάρος των υπόπτων. Εδώ όμως εμείς πρέπει να αλλάξουμε τον νόμο για τον κύριο Ετέν. Μπορούμε να έχουμε αντίγραφα των διαφανειών σας γιατί είπατε πάρα πολλά πράγματα αλλά τα είπατε πολύ γρήγορα. Και θα ήθελα να μάθω τι δεν πάει καλά όχι μέσα στη δική σας υπηρεσία αλλά με την Europol κτλ υπάρχουν τεράστιες εγκληματικές δραστηριότητες και δεν καταφέρνουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Τι δεν πάει καλά λοιπόν. Έλλειψη πόρων ή απαιτείται να υπάρξει ένα επιπλέον ομοσπονδιακό επίπεδο γιατί έχουμε πάρα πολλά κράτη-μέλη πλέον. Και τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεστε, τι θα πρέπει να συστήσουμε εμείς στην έκθεσή μας το επόμενο έτος για να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Σόντεργκάρντα. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες σας. Θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι δεν θα μου δοθούν οι απαντήσεις. Θα τις θέσω παρόλα αυτά. Εγώ θα ήθελα να μάθω ποια είναι πραγματικά η πραγματική η ουσιαστική εμβέλεια της κυβερνοεγκληματικότητας. Όταν μιλάμε για λαθρεμπόριο τσιγάρων, σαν παράδειγμα, γνωρίζουμε με τι, και για, τι ποσότητες μιλάμε. Έχουμε τέτοιου είδους δυνατότητα ποσοτικής καταμέτρησης ε, του οργανωμένου εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και μάλλον τον κυβερνοχώρο γενικότερα. Ε, το οργανωμένο έγκλημα τι ακριβώς ε, ρόλο παίζει, ποιο είναι το ποσοστό του στο στο εγκλήμα του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, θα ήθελα να κάνω επίσης και μία επιπλέον παρατήρηση. Κάθε μορφή εγκληματικότητας έχει σαν βαστικό στόχο τον πλουτισμό. Και αυτό σημαίνει ότι ε, κάποιοι θα βγάλουν λεφτά από αυτήν την ιστορία. Όταν λοιπόν μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συλλάβουμε τους ε, κυβερνοεγκληματίες, στην ουσία θα πρέπει να βρούμε ε, τον σωστό τρόπο που επιτρέπει σε κάποιες ε, ποσότητες χρημάτων σημαντικές να φεύγουν από αυτό που ονομάζουμε κανονικές παραδοσιακές εμπορικές δραστηριότητες. Και όταν προσπαθούμε να σταματήσουμε το κυβερνοέγκλημα η ουσία της προσπάθειας είναι να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των χρημάτων που κυκλοφορούν. Και εδώ ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως. Πώς θα μπορέσουμε να μάθουμε ποιος ωφελείται από την εγκληματική δραστηριότητα. Αυτά είναι θέματα τα οποία λοιπόν τα οποία καταλήγουν στο ότι στόχος της εγκληματικότητας είναι το να βγάλουν κάποιοι χρήματα και αυτά τα χρήματα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε σε ποιους πηγαίνουν και ποιους ωφελούν. Κυρία Φαϊό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους τρεις ομιλητές, θα συμφωνήσω μαζί τους ότι αυτά τα οποία ακούσαμε μας δημιουργούν ορισμένα προβλήματα. Το έγκλημα αυξάνεται ε, σε καθημερινή βάση, νέα θέματα τίθενται και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε προς τα πού θα πάει η τεχνολογική πρόοδος. Παραδέχεστε κι εσείς ε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης ασφάλεια στο διαδίκτυο, είμαστε πάντα ένα βήμα πίσω. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι βέβαια χρησιμοποιούν τον διαδίκτυο, ψωνίζουν online, έχουν ε, πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και σε πάρα πολλά πεδία, σαν παράδειγμα στα κοινωνικά δίκτυα, δεν υπάρχουν δυνατότητες ε, πραγματικού ελέγχου και έτσι έχουμε εγκαταλείψει τους πολίτες και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν φαίνεται ότι έτσι θα αντιμετωπίσει η Ένωση το κυβέρνο έγκλημα. Είπατε όμως ότι δεν θα υπάρξουν επικαλύψεις ανάμεσα στους οργανισμούς, αλλά είπατε ότι και εσείς από μόνοι σας δεν μπορείτε να παρέχετε πλήρη εκάλυψη και ασφάλεια. Πώς θα μπορούσατε λοιπόν να χρηματοδοτήσετε την καταπολέμηση του εγκλήματος από πού θα προέλθουν τα επιπλέον ποσά τα οποία απαιτούνται, εμείς ζούμε μια πολύ σοβαρή οικονομική και πιστοτική κρίση και έχουμε δυσκολία να βρούμε τα οικονομικά μέσα που θα μας επιτρέψουν να βρούμε νέα τεχνολογικά μέσα. Δεν έχουμε χρήματα για μελέτες, έχετε κάποια συγκριτικά δεδομένα ανάμεσα στις διάφορες χώρες της Ένωσης, υπάρχουν κάποιες καλές πρακτικές, υπάρχουν κάποια παραδείγματα από το παρελθόν τα οποία είναι επιτυχή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου. φτάνουμε στους ε, συντονιστές. Ο και έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους τρεις προηγούμενους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τις οποίες έκαναν. Οι ομιλίες τους ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, ιδιαίτερα γιατί τον τελευταίο χρόνο ήμουν σκιώδης εισηγητής για τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιθέσεις στα, στα συστήματα πληροφορικής. Υπάρχει ένα θέμα πολύ σημαντικό στην οδηγία αυτή, η εναρμόνιση των ποινών που εφαρμόζονται, που είναι εφαρμοστές καλύτερα ε, στους κυβερνοεγκληματίες πέρα από το επίπεδο της επιβολής των ποινών μας ανησύχησε το γεγονός το ότι οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές συναντούν πάρα πολλές δυσκολίες στην διατήρηση του σωστού ρυθμού αντιμετώπισης του προβλήματος γιατί οι τεχνολογίες αναπτύσσονται συνεχώς και οι παρανομίες επίσης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τις δικαστικές αυτές αρχές στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν νόμοι οι οποίοι ε, τιμωρούν αυτούς τους παρανόμους. Οι νόμοι αυτοί, όπως είπε όμως και η κυρία Κεμενέρ, δεν εφαρμόζονται με τον σωστό τρόπο και αυτό γίνεται γιατί οι αρχές που είναι υπεύθυνε για την επιβολή αυτών των νόμων δεν έχουν τη σωστή κατάρτιση και ενημέρωση. Στα πλαίσια αυτής λοιπόν της νέας οδηγίας ενθαρρύνουμε την κατάρτιση των δικαστών στον τομέα της εγκληματικότητας στον κυβέρνοχώρο. Χαίρομαι λοιπόν που ξεκίνησαν και στη Γαλλία κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες. Αλλά οι προσπάθειες αυτές κατάρτισης θα μπορούσαν να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί το κυβέρνο έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα. Όπως είπατε πολύ σωστά, αυτή η δραστηριότητα διαπράτεται σε όλες τις χώρες του κόσμου και από παντού. Ένα πράγμα θα προσθέσω ακόμα για την κυρία Κεμενέρη, η οποία το είπε άλλωστε. Δεν έχουμε σωστό ορισμό αυτής της μορφής της εγκληματικότητας. Χάρηκα που σας άκουσα να λέτε κάτι τέτοιο γιατί εμείς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που είχαμε με το Συμβούλιο συναντήσαμε από πλευράς του Συμβουλίου πάρα πολλές αντιστάσεις για την προσπάθειά μας, την προσπάθειά μας εισαγωγής ορισμών και ε, ε, ε, ε, καλυπτόμενο πίσω από την επικουρικότητα το Συμβούλιο δεν θέλησε να προχωρήσει. Λοιπόν, σχετικά τώρα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξει πλήρης προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ανεξαρτήτως των ιστοσελίδων τις οποίες χρησιμοποιούμε, κάθε τέτοια σελίδα ζητά να υπάρξουν προσωπικά δεδομένα και είναι δύσκολο να τα παρακολουθήσει κανείς από κοντά όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάλμπρικ τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ε, τρεις ομιλητές για τις ε, καλές παρουσιάσεις τους. Θα ήθελα να σας πω εξ αρχής ε, ότι εγώ είμαι υπέρ της δημιουργίας αυτού του νέου κέντρου της Σα Σας εύχομαι καλή τύχη στα νέα σας καθήκοντα και νομίζω ότι τα καθήκοντα που αφορούν ε, και την ε, πρόληψη αλλά και την κατάρτιση έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί ουσιαστικά και η αστυνομία νομίζω ότι όντως θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα όμω να σχολιάσω τον ορισμό του κυβερνοεγκλήματο που αναφέρθηκε στην αρχή. Ο ορισμό αυτό είναι κάπω ασαφή. Θα ήθελα να πω εγώ με σαφήνεια δεν είναι λίγο ασαφή. Είναι εντελώ ασαφή και από νομική σκοπιά είναι απαράδεκτο να συζητούμε σε επίπεδο πολιτικής και για ένα ουσιαστικό σημαντικό ποινικό ζήτημα χωρίς να έχουμε ένα σαφή ορισμό περί τίνος πρόκειται για να ε, βάλουμε το διαδίκτυο ή τον κυβερνοχώρο σε ένα κουτί που λέγεται έγκλημα στον κυβερνοχώρο δεν είναι μια νομική προσέγγιση αυτή. Θα πρέπει να έχουμε κάτι που να είναι σαφές στο κοινό και στους νομικούς και στους δικαστές. Δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό, αλλά θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς. Και νομίζω ότι η δουλειά που κάναμε σε ό,τι αφορά την οδηγία για την πρόσβαση στα συστήματα πληροφορικής, ε, όπου αναφερόμαστε σε εγκλήματα που άμεσα σχετίζονται με συστήματα πληροφορικής, αυτή είναι μια προσέγγιση που εγώ θεωρώ ότι είναι πιθανό να ακολουθήσουμε. Εξακολουθώ να βλέπω προβλήματα εκεί σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Τώρα να βάζουμε τα πάντα ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πάτη, παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησία ε, μέσα σε ένα κουτί, γιατί όλα αυτά είναι στο διαδίκτυο και να τα αποκαλούμε έγκλημα στον κυβερνοχώρο δεν είναι ο τρόπο τρόπο να αντιμετωπίσουμε, γιατί αυτά τα εγκλήματα είναι εγκλήματα που ήδη τα γνωρίζουμε και ήδη τα ρυθμίζουμε, τα έχουμε ρυθμίζει και τα έχουμε στου ποινικού μα κώδικε και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όπω στον κανονικό κόσμο, στο μη ψηφιακό κόσμο, όταν έχετε σύνδεση με το ψηφιακό κόσμο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε και με τις ερευνητικές μεθόδους. Βεβαίως και θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Αλλά κύριε Ντίας Δεμέρα, αναφέρατε την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ προστασίας των δεδομένων και της έρευνας. Είδαμε ήδη αυτή τη συζήτηση σχετικά με την εξέβρεση ισορροπίας ε, μεταξύ του σεβασμού των ελευθεριών και της ασφάλειας αλλά να σας πω ότι έχουμε κάποιες αρχές κράτους δικαίου και έχουμε θεμελιώδη δικαιώματα και κάθε εισβολή, κάθε ερευνητικό μέτρο θα πρέπει να αιτιολογείται από νομική σκοπιά. Όχι μόνο δηλαδή να θεωρείται ότι έχει νόημα πολιτική σκοπιά η βοήθα, αλλά θα πρέπει να αιτιολογείται από νομική σκοπιά ω απολύτω απαραίτητο σε μια δημοκρατική κοινωνία και ότι είναι αναλογικό προκειμένου να ε, πετύχει το στόχο όσων έχουμε συμφωνήσει. Και εδώ συμφωνώ μας, είπε ο κύριος χρειαζόμαστε έρευνα και χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα κάνουν καλές έρευνες, όχι μόνο μέτρα εποπτείας, παρακολούθησης και βάσεις δεδομένων. Πρέπει να ανταλλάξουμε βέλτιστα παραδείγματα ερευνητικών μέτρων και να επικεντρωνόμαστε σε υπόπτους, όχι σε αγνώστους. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Να κλείσουμε με τον κύριο Μάλντερ. Ευχαριστώ. Δεν μπόρεσα να ακούσω όλες ε, τις παρεμβάσεις, παρά μόνο τις τελευταίες. Και ακούγοντας τους τελευταίους ομιλητές, ε, μου ήρθε στο νου το εξή. Ε, εγώ ε, πραγματικά είχα αναφερθεί και είχα αναφέρει πόσο λυπάμαι για την απουσία ενός Ευρωπαίου εισαγγελέα. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερο ευρωπαϊκό συντονισμό. Και ε, το, το προβλέπει η συνθήκη, αλλά μέχρι τώρα κάποια κράτη-μέλη είναι κατά αυτού του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. λοιπόν, ε, τι πιστεύει το πάνελ σχετικά με το θέμα αυτό. Όπω, ε, ε, σας είπα, έλειπα κατά το πρώτο τμήμα και θα πρέπει να φύγω και σε λίγο για άλλη συνεδρίαση, αλλά σίγουρα ε, οι βοηθοί μου θα σημειώσουν τι απαντήσει σα. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσουμε στους προκεκλημένους μας ε, τη δυνατότητα να απαντήσουν και πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το συγκεκριμένο κλάστερ μέχρι τις 5.30. Έχετε 5 λεπτά, να ξεκινήσουμε από την κυρία Κεμένερ. Σας ευχαριστώ. Να κάνω κάποιες διευκρινήσεις ε, για τα σχόλια και τις ερωτήσεις που ακούστηκαν. Κυρίως ε, σε ποινικό θέμα από την αρχή της συζήτηση ε, αναφέρουμε αυτό το θέμα του ορισμού. Είναι σημαντικό και αυτό όταν μιλάμε για έγκλημα στον κυβερνοχώρο, μου φαίνεται απολύτως απαραίτητο. Τώρα η ερώτηση για την αξιολόγηση των φαινομένων. Ναι, βέβαια. Είπατε εξ αρχής ότι δεν υπάρχει απάντηση. Είναι μία από τις δυσκολίες. Έχουμε πολλά εργαλεία πολλές εκθέσεις ε, στον ιδιωτικό τομέα, αλλά καμία έκθεση στα χέρια των δημοσίων αρχών. Τουλάχιστον αυτό ισχύει στην Γαλλία υπήρξε ένα ειδικό φάκελο ε, μία έκθεση ε, του ειδικού παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της εγκληματικότητα, ε, όπου αναφερόταν στην χαρτογράφηση του φαινομένου, όμως δεν μπορούμε να πούμε σήμερα πώς, ποιο ακριβώ είναι το ποσοστό του οργανωμένου εγκλήματο που δραστηριοποιείται στον κυβερνό χώρο. Είναι σημαντικό να έχουμε βέβαια αυτά τα αριθμητικά στοιχεία και δημόσια συμφωνώ σε ό,τι αφορά ε, τις υποκλοπές. Αναφέρθηκε και αυτό. Στη Γαλλία ισχύει ε, δεν προβλέπονται από τα κειμενά γιατί μπορούμε να κάνουμε κάποιες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και να τις μεταφέρουμε και στο διαδίκτυο. Αλλά φυσικά υπό έλεγχο δικαστικού ε, και Ξέρετε ότι το τελευταίο έτος ε, κατόπιν της νομοθεσίας που έχουμε για την πρόληψη και για την τήρηση της εσωτερικής ασφάλειας ε, μπορεί να γίνει αυτή η παρακολούθηση, αυτές ε, οι παρακολουθήσεις ε, μπορεί να γίνουν ε, σε ό,τι αφορά τον όγκο των δεδομένων, τα δεδομένα δηλαδή που κυκλοφορούν και όχι ως προς το περιεχόμενο των δεδομένων και να διαρκέσουν ένα μήνα. Έχουμε στη Γαλλία βέβαια ακόμη ένα κενό. Ουσιαστικά γίνονται κάποιες πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα προσωπικές και εγώ μπορώ να σας πω ότι παράλληλα έχω και διοικητικές δραστηριότητες ε, και δεν έχω ακόμη μία θέση, δεν ασχολούμαι δηλαδή αποκλειστικά με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, ενώ θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάποιες θέσεις ε, στο επίπεδο κεντρικής διοίκησης, ε, κάποιος που ασχολείται και με το ψηφιακά. Έτσι λοιπόν αυτή η ειδική ερευνητική υπηρεσία ε, υπάρχει εγώ νομίζω στο δικαστικό επίπεδο θα πρέπει επίσης να ακολουθήσουμε αυτή την εξειδικευσή μου φαίνεται θεμελιώδες και σημείωσε επίσης και την ανάγκη κατάρτισης ε, σε διεθνές επίπεδο, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Παραδείγματο χάρη έχουμε μια πολυτομιακή σχολή ε, σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των δικαστών στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος ε, και ε, σημείωσα επίσης ότι θα παρουσιάσετε τις δραστηριότητες του κέντρου και αυτό δυστυχώς δεν είναι ακόμη γνωστό σε πολλούς δικαστικούς και είναι κρίμα. Θα αναφερθώ και στο θέμα της χρηματοδότησης. Νομίζω ότι και εδώ μια συνεργασία δημόσιο-ιδιωτικού τομέα θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Συχνά έχουμε τους ιδιώτες που προτείνουν ε, προγράμματα κατάρτισης και στους δικαστές και στους εισαγγελείς, αλλά πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Νομίζω ότι τα κράτη δεν θα πρέπει ε, να υποχωρήσουν στην κατάρτιση αυτή Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κονδύλια και από τον ιδιωτικό και από το δημόσιο τομέα για να βελτιωθεί αυτή η κατάρτιση, η οποία θα πρέπει να είναι πολυτομεακή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα σε διεθνέ επίπεδο, γιατί τελικά όλοι στην ίδια κατάσταση βρισκόμαστε, αν μπορώ να το πω έτσι. Δεν ε, ξέρω αν αναφέρθηκα σε όλα. Αναφερθήκατε νομίζω και στο τραπεζικό απόρριτο και την πρέπει και εκεί να υπάρξει εξέβρεση ισορροπίας Κοιτάξτε, δεν έχουμε χρόνο. Μία από τις δυσκολίες ε, είναι η ανάπτυξη ε, δράσεων. Ε, έχουμε, παραδείγματο χάρη, κάποιους τρόπους όπως οι προπληρωμένες κάρτες που επιτρέπουν να μην μπει κανείς καθόλου να μην χρησιμοποιήσει το τραπεζικό σύστημα. και ε, επίσης αναφερθήκαμε και στην κατάσχεση του πραγματικού χρήματος και τι, τι κάνουν. Ε, οι εγκληματίες θέλουν να κερδίσουν εύκολα χρήματα. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον μηχανισμό, δηλαδή την κατάσχεση ε, των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να βρίσκουμε και σε ποιον ανήκουν αυτά τα χρήματα, όμως νομίζω ότι ε, η κατάσχεση αυτή των περιουσιακών στοιχείων είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση του κλίματος στον κυβερνοχώρο. Ευχαριστώ. Ε, και εγώ δεν θα ξεπεράσω τα πέντε μου λεφτά και σας το υπόσχομαι. Νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να καταρτιστεί το σύστημα και μετά να το αξιολογήσουμε σε ένα χρόνο. Ε, δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιολογήσουμε αν χρειαζόμαστε έναν Ευρωπαίο εισαγγελέα. Ε, θα δούμε αν μπορούμε τουλάχιστον θα έχουμε κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός. Επίσης λυπούμε που σας το λέω, αλλά όταν ε, ε, καλούμε στην ε, Europol άτομα για σημαντικές έρευνες, οι μισοί δεν έρχονται γιατί οι χώρες τους δεν έχουν χρήματα για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα πρέπει να πληρώνουμε τουλάχιστον τις πτήσεις σε οικονομία αεροπορική θέση για να μπορέσουμε να συλλέξουμε τα στοιχεία. Επίσης υπάρχουν υπάρχουν διάφοροι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών. Εδώ έχετε διάφορες. Τώρα όμως χρειάζονται χρήματα. 25 ευρώ αναδιεύθυνση ε, ηλεκτρονική. Εάν αυτά τα έξοδα όμως ποιος θα τα αναλάβει η χώρα που έχει το δικαστικό σύστημα που παρακολουθεί τους ε, ε, ηλεκτρονικούς παρόχους ή ποιος. Ορισμένες χώρες δεν μπορούν είτε να αντέξουν το κόστος ή δεν θέλουν να ε, πληρώσουν. Οπότε εμάς τελείωσαν τα χρήματά μας και δεν έχουμε τώρα χρήματα για το κέντρο πάταξης ε, ε, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι ε, υπολογισμοί για το κόστος για το κυβερνοέγκλημα και πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το όφελος και τι θα κοστίσει. Και βεβαίως δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος επενδύσεων και εξόδων και δεν θα θα καταπολεμήσετε ε, το κυβερνοέγκλημα με το ε, να αυξήσετε την προστασία αλλά πλούστατα με το να γίνει πολύ δαπανηρή η ποινή ε, εάν σας πιάσουν. Υπάρχουν διάφορες εγκληματικές πράξεις διαφόρων ομάδων αλλά γενικώ νομίζω ότι οι συμβουλή ήταν πολύ καλές αλλά το βασικό είναι πόσο γρήγορα θα χρηματοδοτηθούμε διότι βλέπουμε ότι ε, εάν κινηθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώσπου να το πιάσουμε έχει μοιραστεί και υπάρχουν χώρες ε, όπου εξαφανίζονται τα χρήματα και όχι μέσα σε χρόνια αλλά μέσα σε μια μέρα και μιλάμε για εκατομμύρια. Είπατε αν ε, θα μπορέσουμε να λύσουμε τα πάντα. Όχι, είμαστε πολύ μικροί και δεν υπάρχει και λόγος η συνολική αντιμετώπιση είναι ότι ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του, εμείς θα βοηθούμε ο ένας τον άλλον, η ΣΥΠΟΛ έχει την Αστυνομική Ακαδημία, θα βοηθήσουμε ε, και για πρώτη φορά αυτά θα μπορέσουν να γίνουν συντονισμένα ώστε ο καθένας να κάνει το δικό του τμήμα συγχρόνως για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουμε πολλά. Χρειαζόμαστε έναν ε, δημόσιο κατήγορο. Έχω μία προσωπική άποψη επ' αυτού, αλλά δεν νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να σας απαντήσω. Ευχαριστώ. Λίγες παρατηρήσεις. Κύριε Ντύρες Ντεμέρα, ξεκινήσατε μιλώντας για την ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής ζωής και ασφαλείας και της καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος. Κάθε φορά που συζητάμε αυτά τα θέματα καταλήγουμε στο ποιο ήταν, ποια θα ήταν η σωστή ισορροπία μεταξύ των αντικρουωμένων συμφερόντων και ουσιαστικά εσείς φοβάστε ότι η πάροχή διαδικτυακών υπηρεσιών ε, θα κρυφτούν πίσω από την προστασία δεδομένων για να μην συνεργαστούν για την πάταξη του κυβερνού εγκλήματος. Ε, νομίζω ότι ε, ε, καλό θα ήταν, όπως είπε και ο Γιάνν Άλμπρεχτ, να συζητήσουμε τα βασικά δικαιώματα και να δούμε αν υπάρχουν μέτρα τα οποία χρειάζονται και πώς ε, θα συνεργαστούμε παραδείγματος χάρη με το κέντρο για το κυβερνοέγκλημα της Europol και να δούμε πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν καλύτερα καθενός τα συμφέροντα και να μην ε, κρυβόμαστε πίσω από άτομα που δεν θέλουν να συνεργαστούν. Ο κύριος Νιούτον Τζον αναφέρθηκε στην παγίδευση στο ε, διαδίκτυο και αυτό δεν απαγορεύεται στον, ε, στην νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αν υπάρχει μία δίσδυση ή Ε, υπάρχει παρακολούθηση των συζητήσεων αυτά θα μπορούν να ε, γραφτούν σε, κάποια, σε κάποιο μέσο να τα ακούσει κάποιος δικαστής και να ελέγξει ουσιαστικά. Είμαστε σε μια κοινωνία όπου παραδείγματος χάρη στις συζητήσεις πολλές φορές η αστυνομία παρακολουθεί τις συνομιλίες αλλά πρέπει να ελέγχεται, πρέπει να ξέρουμε τι έγινε διαφορετικά. Όντως κινδυνεύουν τα βασικά μας δικαιώματα. Πολλά πρέπει να γίνουν, αλλά είτε υπό την προστασία της δικαστικής αρχής ή της αρχής προστασίας δεδομένων ή και των δύο. Ένα άλλο βασικό θέμα ήταν το σχόλιο του κυρίου Εντσού, ο οποίος είπε ότι ούτως ή άλλως ε, δεν έχετε ιδιωτική ζωή στο διαδίκτυο. Μην συγχαίετε διαφορετικά πράγματα. Είμαι πεπισμένος ότι στο διαδίκτυο Ε, ε, έχουμε πάρα πολλά ε, λέσεις στο που ζητούν πολλά προσωπικά στοιχεία που δεν χρειάζονται. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα. Απλώς και μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες πληροφορίες δεν αποκλείει το ότι ε, ε, θα έπρεπε να παραδώσουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τα δεδομένα. Όχι. Θα βρεθεί μία μέση οδός και ελπίζω ότι θα πετύχουμε. Πολλοί μίλησαν για σαφείς ορισμούς, για ε, νομική ασφάλεια, νομική ασφάλεια και σαφείς ορισμοί και ε, εναρμονισμένη προσέγγιση σε όλη την Ευρώπη είναι προ συμφέρον όλων που καλύπτουν αυτό το χώρο είτε για την προστασία των δεδομένων είτε σαν διοκτικές αρχές και θα έπρεπε να βοηθηθούμε για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Το εάν ο υπεύθυνο θα έπρεπε να είναι ο δημόσιος εισαγγελέα, ε, θα το αφήσω στη διάκριση του κοινού. Ευχαριστώ λοιπόν και τους τρεις εισηγητές γιατί μπόρεσαν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ασχοληθούν με ένα θέμα το οποίο θα έλεγα θέτει πάρα πολλά νέα προβλήματα και νέα πεδία προβλημάτων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε γιατί στο διαδίκτυο υπάρχουν πάντα εκατομμύρια πολίτες και ιδιαίτερα παιδιά και στην ουσία παραμένουν απροστάτευτα. Λοιπόν, είναι σαφές ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τα περιθώρια δράσης αυτών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να βλάψουν τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσίασή σας. Κλείσαμε λοιπόν με το δεύτερο γύρο. Εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος στο στήσιμο αγώνων και στη διαφθορά στα σπόρα. Θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Δημοσθένη Χρυσικό από το UNODC. Και μετά θα ακούσουμε την κυρία Εμινέ Μποσκούρτ, η οποία είναι η συγγήτρια. Η συζήτηση θα γίνει όπως συνήθως, δηλαδή ε, δύο λεπτά για τον καθένα από εσά και μετά ε, θα ακούσουμε και τις ερωτήσεις των συναδέλφων. 15 λεπτά λοιπόν έχει το λόγο ο κύριος Χρυσικός. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές. Θα ήθελα και εγώ να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την πρόσκλησή σας έτσι ώστε να παρακολουθήσω τη συνεδρίασή σας εξ ονόματος της Υπηρεσίας των Ηνωμένων ε, Εθνών για τα Ναρκωτικά και το έγκλημα. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν και τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σήμερα και αύριο. Τώρα, η βάση και ο στόχος της παρουσίασής μου σήμερα το απόγευμα είναι τα προβλήματα, ή προκλήσεις οι οποίες τίθενται από την παράνομη χρήση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των αθλητικών αγώνων και το στήσιμο το λεγόμενο των αγώνων αυτών και η προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών για να καταπολεμηθεί αυτή η μορφή εγκληματικότητας. Πριν εξετάσουμε λοιπόν τις προοπτικές της UNODC, της Υπηρεσίας λοιπόν για τα Ναρκωτικά των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να πούμε ότι το φαινόμενο αυτό είναι κάτι το οποίο συναντάμε όλο και περισσότερο και προσπαθούμε να δούμε αν οι απαντήσεις μέσω της ε, νομοθετικής οδού είναι απαραίτητες και αν είναι οι καλύτερες. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αποδείξεις όλο και περισσότερο ότι ο αθλητισμός ε, δεν είναι άτρωτος από το ε, στήσιμο των αγώνων, το φαινόμενο του στήσιματος των αγώνων και της καταχρηστικής χρήσης των αθλητικών δραστηριοτήτων υπάρχει θα έλεγα ένα σύνολο ε, ε, μέσων που χρησιμοποιούνται για την, την εγκληματική ε, χρήση των αγώνων των αθλητικών. Αυξάνεται ο αριθμός των στημένων αγώνων και αυτό εξηγείται εν μέρη από την αύξηση των προσφορών σε επίπεδο στοιχημάτων online, κάτι το οποίο με τη σειρά του έχει αυξήσει θα έλεγα τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν άμεσα οικονομικά συμφέροντα σε σχέση με τις αθλητικές δραστηριότητες. Αυτό είναι κάτι που ξεπερνά λοιπόν τα εθνικά σύνορα, τα στοιχήματα αυτά μέσω του διαδικτύου. Είναι κάτι το οποίο θα έλεγα περιορίζει και τις δυνατότητες σύλληψης των ε, δραστών αν και συγκεντρώνουμε την προσοχή μας κυρίως στις προηγούμενες συναντήσεις και σε επίπεδο ορολογίας, παρενθετικά μόνο θα ήθελα να σας θυμίσω τον ορισμό ο οποίος χρησιμοποιείται σε μια πολύ πρόσφατη μελέτη η οποία έγινε για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, μια γεωγραφική παρουσίαση θα έλεγα των ρυθμίσεων των νομικών σε σχέση με το στήσιμο των αγώνων. Δίδεται λοιπόν η εξής θα έλεγα μορφή ορισμού που χρησιμοποιείται και από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η εκμετάλλευση καταχρηστική των αποτελεσμάτων των αγώνων καλύπτει το σύνολο των αθλητικών δραστηριοτήτων, αγώνες ε, πολλών μορφών, έτσι ώστε να ε, υπάρξει οικονομικό όφελος για τον δράστη ή για άλλους, και να μην υπάρχει η αβεβαιότητα η οποία χαρακτηρίζει γενικά τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου αγώνα. Η ανάγκη λοιπόν καταπολέμησης του στισίματος των αγώνων είναι κάτι το οποίο για μας καθορίζεται από διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι το φαινόμενο αυτό είναι κοινωνικού ενδιαφέροντος, είναι κάτι το οποίο θίγει τις πνευματικές και πολιτιστικές αξίες του αθλητισμού και θέτει να αμφισβητήσει και τον οικονομικό ρόλο του αθλητισμού. Αναγνωρίζοντας λοιπόν το δημόσιο συμφέρον εδώ, έχει σημασία να προσπαθήσουμε να δούμε αν τα μέτρα μέσω των ποινικών διώξεων είναι επαρκή για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που δημιουργούνται από το στήσιμο των αγώνων. Υπάρχουν αρκετές θα έλεγα αποδείξεις που δείχνουν ότι η καταχρηστική ε, θα έλεγα χρήση των αποτελεσμάτων δεν είναι μόνο κάτι που παραβιάζει τους αθλητικούς κανόνες αλλά φύγει το κοινό γενικότερα. Στον τομέα του ντόπινγκ σαν παράδειγμα η χρήση των μηχανισμών της ποινική δικαιοσύνης μπορεί να βοηθήσει την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ε, ο χαρακτηρισμός αν είναι θα έλεγα ένα γενικότερο τύπου, μια γενικότερου τύπου ε, εγκληματική δράση ή μια πιο συγκεκριμένη εγκληματική δράση η οποία θα έλεγα ορίζεται με ξεχωριστό τρόπο και εμπλέκει αποκλειστικά αθλητικές δραστηριότητες είναι κάτι το οποίο φύγει φυσικά και τους εμπλεκομένους στις αθλητικές δραστηριότητες, προκαλεί φαινόμενα διαφθοράς και κάτι τέτοιο φυσικά είναι ποινικά κολάσιμο. Η έκφραση στήσιμο αγώνων αντικαθίσταται μερικές φορές το match ε, fixing από δωροδοκία αθλητικού τύπου. Αυτό δείχνει ότι οι αθλητικές δραστηριότητες ε, επηρεάζονται από τη διαφθορά. Ε, σε επίπεδο οργανωμένου εγκλήματος τα προβλήματα που δημιουργούνται με τα στοιχήματα είναι γνωστά, αλλά έχουμε φτάσει σε νέα επίπεδα περιπλοκότητας με πάρα πολλούς εμπλεκομένους σε πάρα πολλές χώρες και σε πολλές φυσικά νομικές δικαιοδοσίες. Υπάρχουν νέες εταιρείες στοιχημάτων offshore και αυτή η περιπλοκότητα υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείται το δίκτυο και από το οργανωμένο έγκλημα με ε, διεθνή πλέον διάσταση. Ένας άλλος ε, παράγοντας ο οποίος καλεί την ποινική δικαιοσύνη είναι η έκπληνση χρήματος, βρώμικου χρήματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο άπτεται και της διαφοράς και πρέπει να εξετάσουμε προσωπικά τα συστήματα έκπληξης χρημάτων ε, στα πλαίσια της, ε, του στισήματος των αποτελεσμάτων των αγώνων. Υπάρχουν βέβαια λόγω των πολλαπλών δικαιοδοσιών ε, πολλές διαφορετικές νομικές ρυθμίσεις και η ενιαία αθλητική αγορά δεν καθορίζεται με ενιαίο τρόπο. Υπάρχουν πολλοί εταίροι και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο που λειτουργούν. Η παροχή πολλές φορές είναι εγκαθεστημένοι σε χώρες οι οποίες έχουν τις αθλητικές δραστηριότητες, αλλά έχουν επίσης την έδρα τους και σε χώρες οι οποίες δεν ελέγχουν τις δραστηριότητες αυτές και είναι πολύ δύσκολο να αναλάβει κανείς νομική δράση εις βάρος των παροχέων οι οποίοι λειτουργούν online δεν υπάρχει διαφάνεια και ακριβώς τα στοιχήματα με αυτόν τον τρόπο καθίστανται κάτι το πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, για τους εγκληματίες και ακριβώς τα αποτελέσματα και τα κέρδη αυτών των δραστηριοτήτων αυξάνουν το ξέπλυμα του χρήματος. Και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη λοιπόν συστηματικότερης ε, νομικής παρέμβασης για την καταπολέμηση των αρνητικών αποτελεσμάτων του συστήματος των αθλητικών αγώνων. Αυτό δεν επηρεάζει ε, τις αθλητικές ε, αρχές να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό μεμονωμένα γιατί τίθεται και θέμα εδώ αθλητικής αυτονομίας και πάρα πολλές φορές ε, οι εισαγγελίε και οι ανακριτικές αρχές συνεργάζονται με τις αθλητικές αρχές χωρίς να υπονομεύουν όσους εμπλέκονται στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας που δεν είναι μόνο αθλητικές αρχές αλλά και επιστοτικοί οργανισμοί κτλ. Υπάρχουν λοιπόν πολλαπλά επίπεδα θα έλεγα νομικής ε, ανταπόκρισης είτε μια μορφή γενικής αντιμετώπισης είτε μια μορφή εξειδικευμένης αντιμετώπισης και αυτό δείχνει ότι έχουμε ένα περιθώριο ευελιξίας εδώ για την αντιμετώπιση του προβλήματος και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε νομικά ποια είναι τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό ακριβώς τα πολυμερή μέσα τα οποία διατίθενται και τα οποία το UNODC θα έλεγα χρησιμοποιεί για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος όπως η Σύμβαση του Παλέρμο του 2002 και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 2005 για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τα μέσα αυτά παρέχουν ε, κατάλληλες θα έλεγα απαντήσεις έτσι ώστε οι εθνικές δικαιοδοσίες να αντιμετωπίζουν το στήσιμο των αγώνων στα πλαίσια της χρήσης της ποινική ε, ε, δικαιοσύνης στήριξης των ένομων μέσων που χρησιμοποιούνται και μέσω ισχυρών αποτελεσματικών μηχανισμών διεθνούς συνεργασίας. Ιδιαίτερα η, διάσκεψη, η σύμβαση του Παλέρμο είναι θα έλεγα ένα βασικό ε, μέσο, σφαιρικό μέσο με 171 χώρες οι οποίες έχουν επικυρώσει τη σύμβαση αυτή και οι περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες επίσης. Η σύμβαση του Παλέρμο λοιπόν δίδει ένα ευρύτατο πεδίο συνεργασίας για την, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος όπως υπάρχει και όπως αναδύεται επίσης και στον τομέα του στισίματος των αγώνων, δίνοντας ευελιξία στους δικαστές της διάφορες χώρες, χρησιμοποιώντας κάποιους ορισμούς όχι για το οργανωμένο έγκλημα, έχουμε ακούσει γι' αυτό, αλλά των εμπλεκομένων στο οργανωμένο έγκλημα, των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων στα πλαίσια σοβαρών εγκληματικών πράξεων. Από την άλλη η, Ευρωπα... Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι το πρώτο ε, ε, έμβικο διεθνές μέσο και δίδει ε, συγκεκριμένες δυνατότητες για την καταπολέμηση του προβλήματος και την ενίσχυση των εθνικών κυρίων κυρίως μέσων για την καταπολέμηση της διαφοράς και την ανάκτηση των σε εισαγωγικά και υπάρχουν όπως είπα πολλές χώρες οι οποίες συμμετέχουν ε, στο μέσο αυτό. Σε επίπεδο ποινική αντιμετώπισης θυμίζω ότι το μέσο αυτό δεν περιλαμβάνει ένα ορισμό της διαφθοράς γιατί θεωρείται κάτι το αρκετά ρευστό. Αντίθετα έχει προτιμηθεί η περιγραφική μέθοδος ορίζοντας κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες είτε με υποχρεωτικό τρόπο είτε με εθελοντικό τρόπο που συνδέονται με κάποιες ε, μορφές διαφθοράς. Για το στήσιμο των αγώνων η υπηρεσία μας ε, προσφέρει πολλές επιλογές για την αντιμετώπιση τους ε, σύμφωνα με τους εξής παράγοντες. Καταρχάς, οι διαπράττοντες σε συγκεκριμένες τέτοιες πράξεις στην περίπτωση κατά την οποία εμπλέκονται και δημόσιοι υπάλληλοι τότε κρατικοί εκπρόσωποι, τότε μπορεί να χρησιμοποιούνται επί τη βάση του άρθρου 50 για τη δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων ή το 15 ή το 19 για την κατάχρηση θέσης. Υπάρχει και ένας δεύτερος παράγον όμως, ανάλογα με τη συγκεκριμένη φύση της εγκληματικής ενέργειας και τον αθλητισμό. Στις περισσότερες χώρες ο αθλητισμός ανήκει στον λεγόμενο ιδιωτικό χώρο αλλά παρόλα αυτά αναλαμβάνεται κυβερνητική δράση συμπληρωματικά και ενισχυτικά της δράσης των αθλητικών οργανωτών. Όπως είπα λοιπόν θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα όρια της εμπλοκής αυτής έτσι ώστε να μην φυγεί η αυτονομία του αθλητικού χώρου. Αντιμετωπίζουμε επίσης και με ποινικέ ενέργειες ε, που έχουν σχέση με την διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα και σε συνεργασία με τη UNODC προβλέπονται και μέσα τα οποία καθορίζουν τους υπευθύνους, τους υπολόγους ανάλογα με τις ευθύνες που έχει αναλάβει σε επίπεδο ποινικό ή σε επίπεδο αστικό. Υπάρχει το θέμα της, του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Εδώ είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται και στον τομέα της, του στισίματος των αγώνων. Υπάρχουν προβλέψεις ε, για την προστασία αυτών που αναφέρουν τα εγκλήματα αυτά ή των, ε, αυτών που δίδουν μαρτυρίες ε, και τέλος λεπτομερές και συγκεκριμένο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου τρόπου αυτού με το οποίο διαπράτεται η εγκληματική αυτή δραστηριότητα καλύπτοντας τη διεθνή της διάσταση. Το UNODC συνεργάζεται επίσης και με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή επί τη βάση ενός μνημονίου συνεργασίας το οποίο υπεγράφει το 2011. Ως εκ τούτου λοιπόν συμμετέχουμε στην δράση της Επιτροπής της Ολυμπιακής για την καταπολέμηση των παρανόμων στοιχημάτων στον αθλητισμό. Ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της ομάδας εργασίας είναι να αντιμετωπιστούν τα θέματα τα οποία άπτονται της νομοθετικής αντιμετώπισης και τα αποτελέσματα αυτής της ομάδας εργασίας οδηγούν σε συγκεκριμένες προτάσεις για την σωστή συνεργασία ανάμεσα στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, το UNODC και άλλες διεθνούς εταίρους επί τη βάση των εμπειριών που έχουμε μέχρι τώρα συλλέξει. Αυτό που έχει ξεκινήσει να γίνεται λοιπόν είναι μια συγκριτική μελέτη για τις ε, προβλέψεις της νομικές για την καταπολέμηση ε, των παρανόμων στοιχημάτων, κάτι το οποίο επεξεργαζόμεθα σε συνεργασία με τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές περιλαμβάνουμε μια συγκριτική μελέτη όλων των τρόπων ποινική αντιμετώπισης του στισίματος των αγώνων και των παρανόμων στοιχημάτων είναι κάτι το οποίο θα ξεπεράσει τις τακτικές ασκήσεις εισαγωγικά που γίνονται στα πλαίσια της συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνοντας τις δυνατότητες συμμετοχής και από άλλες χώρες του κόσμου. Η μελέτη θα μελετήσει επίσης και τις πλευρές οργανωμένου εγκλήματος σε σχέση με το στήσιμο των αγώνων και επίσης θα δώσει επιλογές στους εμπλεκομένους για την δυνατότητα βελτίωσης της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση του φαινομένου χρησιμοποιώντας τα διεθνή μέσα όπως το UNOCT και το UNCA. Και τέλος, θα υπάρξουν και συγκεκριμένα σενάρια αντιμετώπισης του των μεθόδων στισήματος αγώνων έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις προσπάθειες αυτού, αυτών οι οποίοι θέλουν να υπάρξει περισσότερη συνεργασία για την καταπολέμηση του εγκλήματος γενικότερα αντιστοίχων εγκληματικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις νομικές απαιτήσεις που ε, ε, είναι σαφείς και δεδομένες σε επίπεδο διεθνών ποινικών διαδικασιών. Μια επιπλέον προσπάθεια που κάνει το UNODC σαν βασικός εταίρος είναι να υποστηρίξει νομοθετικές προσπάθειες για τον καθορισμό των ποινικών, ε, των ποινικών διαδικασιών υπάρχει και μια παράλληλη διαδικασία για τη δημιουργία ενός μέσου ε, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενός νέου διεθνούς μέσου για ε, το στήσιμο ε, των αγώνων και στοιχημάτων, είναι κάτι το οποίο θα έχει σαν κύριο στόχο τα προληπτικά μέτρα και όχι την καταπολέμηση του φαινομένου. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για περισσότερες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε. Εγώ πιστεύω ότι ο αθλητισμός και ιδίω το ποδόσφαιρο είναι σημείο αναφοράς ε, για πάρα πολλούς νέους. Ότι οι ποινές θα πρέπει να είναι παραδειγματικές. Γιατί υπήρξε ουσιαστικά κάποια έλλειψη βούλησης, ε, κάποια επιφανειακή προσέγγιση σε αυτή την ε, σε αυτό το τομέα, ενώ ο αθλητισμός ε, είναι κάτι που εμπνέει τους νέους, ιδιαίτερα στη χώρα μου. Ε, αυτή τη στιγμή γίνεται πραγματικά σεισμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, και στους δικαστικούς κύκλους, γιατί, ξέρετε, υπάρχουν στημένοι αγώνες στο πρωτάθλημα και έχω την εντύπωση ότι αυτό αντιμετωπίζουν κάποιοι ω ε, κάτι που δεν είναι και πάρα πολύ σοβαρό, είναι κάτι που μα διασκεδάζει. όμω γύρω από αυτό γυρίζουν εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ και οι νέοι μα θα παρακολουθούν όλα αυτά και νομίζουν ότι αυτά είναι τα σημεία αναφοράς. Έτσι λοιπόν εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε παραδείγματικέ ποινέ. γιατί πραγματικά αυτή η υπερβολική αυτή η υπερβολικά επιπόλη προσέγγιση μπορεί να δώσει ένα χειριστό παράδειγμα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο την κυρία Εμινέ Μποσκούρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα ρίξουμε ένα φως στο να βρούμε μια νέα προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά και το στήσιμο των αγώνων στον αθλητισμό Συσυγήτρια για την ευρωπαϊκή διάσταση ε, στον αθλητισμό με την Επιτροπή Πολιτικών Ευθεριών παρουσίασε μια έκθεση για την καταπολέμηση των στημένων αγώνων πέρσι τον Οκτώβριο που ομόφωνα υποστηρίχθηκε από όλα τα μέλη από όλες τις πολιτικές ομάδες από όλα τα πολιτικά κόμματα. Όμω δυστυχώ πέρασε ένα χρόνο και δεν έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδο ε, κατά ε, τη διαφθορά στον αθλητισμό και των στιμένων αγώνων σήμερα. Και πάλι θα μιλήσω για του στιμένου αγώνε εδώ ενώπιον τη Επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και νομίζω ότι σε πολύ σωστή χρονική στιγμή αναφερόμαστε στο θέμα αυτό γιατί όχι μόνο ασχολούμαστε με την έκθεση αυτή, αλλά και αυτή την εβδομάδα θα υπάρχει άτυπο Συμβούλιο Υπουργών στην Κύπρο, υπό την Κυπριακή Προεδρία, που πιθανά θα δημοσιεύσει και μια δήλωση για τους τιμένους αγώνες. Έτσι νομίζω ότι είναι πολύ καλό να δράξουμε αυτή την ευκαιρία για να παράσχουμε και κάποιες συστάσεις ε, στους αρμόδιους υπουργούς αθλητισμού. Όπως είπατε Πρόεδρε, το στήσιμο των αγώνων μπορεί να φαίνεται ως σημασία θέμα, αλλά είναι σοβαρό πρόβλημα στην Ευρώπη. Είναι ένα κερδοσκοπικό έγκλημα με υψηλά έσοδα και χαμηλές ε, ποινές και πολύ χαμηλά ποσοστά εντοπισμού και πολύ συχνά χρησιμοποιείται ως εργαλείο των εγκληματικών ομάδων για την ομοποίηση παρανόμων εσόδων. Ε, ο αθλητισμός ε, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και ε, μια επιχείρηση όπου διακινούνται δισεκατομμύρια ευρώ από τα στοιχήματα, τα δικαιώματα της τηλεόρασης και άλλα και όπου εμπλέκονται τόσα πολλά χρήματα με περιορισμένο έλεγχο από τις δημόσιες αρχές υπάρχει μόνιμος κίνδυνος διαφθοράς, ιδίως λόγω της αύξησης, ε, λόγω της διάδοσης ε, του διαδικτύου. Ε, τα στοιχήματα στο διαδίκτυο φαίνεται να αυξάνονται. Αν δείτε τις στατιστικές από το AIDS του ΟΟΟΥ τα τελευταία χρόνια από 16,3 3 ε, εκατομμύρια ευρώ το 2004 φτάσαμε στα 50,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012. Αυτός είναι ο όγκος ε, των ε, στοιχημάτων, των νόμιμης αγοράς των στοιχημάτων στον αθλητισμό. Δεν υπάρχουν φυσικά νούμερα για την παράνομη αγορά που απειλεί ακόμη περισσότερο την ε, ακαιρεότητα του αθλητισμού καθώς υπάρχουν άμεση συνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Αν δούμε στα κράτη-μέλη μέχρι τώρα, σε 19 από τα 27 κράτη-μέλη και σε 4 υποψήφιες χώρες έχουν ανοιχνευτεί στημένοι αγώνες ε, και έχουν γίνει έρευνες είτε από ενώσεις αθλητικές ή από τις δημόσιες αρχές σε ορισμένες περιπτώσεις όταν ε, η ευρεία πλειοψηφία των κρατών ε, μελών θίγεται από το στημένους αγώνες, ε, βλέπουμε φυσικά ένα πρόβλημα διασυνοριακό, είναι προφανές. Τι βλέπουμε σήμερα, ότι πολλές πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται από πολλούς πρωταγωνιστές προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση, για να αναφέρω κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες Έχουμε από τις ε, αθλητικές οργανώσεις, η UEFA έχει διορίσει 53 αξιωματούχους ε, σε, σε εθνικές ενώσεις. Επίσης και η FIFA ε, έχει σύστημα εγκύρισης προειδοποίησης για την παρακολούθηση πάτων στοιχημάτων. Επίσης και η UEFA είναι στη διαδικασία συστάσεις μνημονίου συνενότησης για να υλοποιήσουν περαιτέρω, για να, περαιτέρω συνεργασία. Η FIFA συνεργάζεται με την Interpol ε, για την ανείχνευση ύποπτων περιπτώσεων. Στα περισσότερα κράτη-μέλη η απάτη στον αθλητισμό θα μπορούσε ε, να υπόκειται στη Γενική Νομοθεσία για τη Διαφθορά. Όμω στα περισσότερα κράτη-μέλη ε, λείπει ένα σχετικό ορισμό για την απάτη στον αθλητισμό στην ποινική νομοθεσία. Και έχω προετοιμάσει ένα έγγραφο το οποίο είναι ιστορικές πληροφορίες για τις συστάσεις. Νομίζω ότι θα μοιραστεί. Το δώσαμε στη γραμματεία. Διαφορετικά θα το βάλουμε εδώ αυτό το έγγραφο έτσι ώστε να μπορούν να το δουν όσο ενδιαφέρονται και θα το στείλουμε και στα μέλη της Επιτροπής σας. Γιατί είναι δύσκολο να σας δώσω όλα τα στοιχεία για όλα τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει αυτή η έλλειψη σε πολλά κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ο πίτροπος για, ε, για τον αθλητισμό συνέστη σε μία ομάδα προκειμένου να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό ε, σχέδιο για τον αθλητισμό. Μισελ Μπαρνιέ ανακοίνωσε ένα σχέδιο δράση για να συζητηθούν τα στοιχήματα και τα τυχερά παιχνίδια στην Ευρώπη και στον αθλητισμό. Ε, Ω ένα από τα κύριε ζητήματα, το Συμβούλιο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή συντάσσει μία σύμβαση ε, και τα κράτη-μέλη θα συμμετάσχουν ε, σε αυτή τη σύμβαση και, μία, και συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες ε, κατά των στιμένων αγώνων. Αυτό που βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από το δημόσιο και από τους κύριους stakeholders, όμως μία συνολική προσέγγιση, μία πλατφόρμα όπου θα έπρεπε να συναντηθούν όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι, τα ενδιαφερόμενα μέρη λείπει. Το Συμβούλιο της Ευρώπης εργάζεται σκληρά για την κατάρτιση της σύμβασης όμως ε, δεν έχει την εξουσία να νομοθετήσει να επιβάλλει κυρώσεις για να στη στημένοι αγώνες ε, στην Ευρώπη ε, χρειάζονται ε, δομές για τη λήψη αποφάσεων. Και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι εξαιρετική πρωτοβουλία, όμως πρέπει να υπάρξει συντονισμό των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει ηγετική θέση και να ακολουθήσει μια προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένου κινδύνου που ανέχονται για τα κράτη-μέλη, ενώ θα λειτουργεί και ω αστιακό σημείο για το συντονισμό μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι μεγάλη γκάμα πρωτοβουλειών ε, που αναλαμβάνονται ε, αλλοσυμπληρώνονται και δεν υπάρχει επικάλυψη. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να τα κάνει αυτά από μόνη της. Όλα τα κυρία διαφερόμενα μέρη διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο να υπάρξει μια καθολική προσέγγιση που να λειτουργεί. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους στισμένους αγώνες στην Ευρώπη αποτελεσματικά. Και προκειμένου να το πετύχουμε αυτό, έχω ε, κάνει κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις ε, στα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη. Οι συστάσεις μου στις αθλητικές οργανώσεις ε, θα ήταν να έχουν μια πολιτική μηδενική συνοχή στη διαφθορά και εσωτερικά και εξωτερικά για να αποτρέψουν τα μέλη των αθλητικών οργανώσεων να δέχονται εξωτερικές πιέσεις. Δεύτερη σύσταση, στις αθλητικές οργανώσεις ε, να δημιουργήσουν ένα κώδικα δεοντολογίας ε, που να καθορίζει τους κίνδυνους που κρύβουν οι στημένοι ακοβοί και να υπάρξουν ε, και κυρώσεις για τέτοιες δραστηριότητες και να υπάρξει και μια απαγόρευση για εταιρείε που προβαίνουν σε παράνομα στοιχήματα. Επίσης, στον κώδικα δεοντολογίας να υπάρξει υποχρέωση για να αναφέρονται οι στημένοι αγώνες και να υπάρχει και ένας μηχανισμός προειδοποίησης επίση να υπάρχει ένα πρόγραμμα για με ξεκάθαρες υποχρεώσεις για του συνδέσμους ε, και τις διάφορες ε, ενώσει και όμως σπονδίες ε, στο Σε Ό,τι αφορά τώρα τις ενώσει, και είναι να υπάρξει μία δεσμευτική συμφωνία μεταξύ όσων δραστηριοποιούνται στο στοίχημα προκειμένου να υπάρξει συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης. Δεύτερον, να δημιουργηθεί μία διαδικασία ε, που θα, ε, ε, όπου οι αθλητικές οργανώσεις θα συνεργάζονται με τις δημόσιες αρχές προκειμένου να ανοιχνεύουν αυτά τα φαινόμενα. Τρίτον, τη συμφωνίες συνεργασίας με κάποιους επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες ε, προκειμένου να εντοπίζονται τα μοντέλα ε, στοιχημάτων. Σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ενορμανισμένη σορισμός των στιμένων αγώνων στο ποινικό δίκαιο και να δημιουργηθεί ένα εργαλείο για την καταπολέμηση των στιμένων αγώνων, να υπάρξει μια συγκεκριμένη μονάδα για την καταπολέμηση των στιμένων αγώνων στα πλαίσια των διοικητικών αρχών, υπάρχει ένας κόμβος συνεργασίας. Τρίτον, ε, να ε, υπάρξει, ε, να υπάρξει δημιουργία κοινών ερευνητικών ομάδων και να υπάρξει συνεργασία των δικαστικών αρχών, των δικαστικών αρχών, να δημιουργηθούν μέσα για την καταπολέμηση των παράνομων ιστοσελίδων, Τώρα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει για το κορολό για να καταπολεμήσει του τιμένου αγώνε, δημιουργώντα μια πλατφόρμα συζήτηση, ανταλλαγή πληροφοριών και των πρακτικών και να συντονίσει τι προσπάθειε των κύριων ενδιαφερομένων μερών, δηλαδή των αθλητικών οργανώσεων, των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στα στοιχήματα, των διοκτικών αρχών κτλ. στην καταπολέμηση των στιμένων αγώνων. Να καταπολεμήσει του στιμένους αγώνε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω συντονισμού των κρατών μελών για να υπάρξει και ένας ορισμός των στημένων αγώνων στο ποινικό δίκαιο. Επίσης, δημιουργία συνεργασίας με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση στοιχημάτων σχετικών με τους στημένους αγώνες. Συμπερασματικά θα έλεγα χρειάζεται μία πλήρης προσέγγιση με τη συνεργασία των αθλητικών οργανώσεων, ε, των διοκτικών αρχών, ε, των δημοσίων αρχών και των ευρωπαϊκών οργάνων. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα για να πολεμήσουμε τους τιμένους αγώνες γιατί το ε, χρωστάμε σε εκατομμύρια Ευρωπαίους για τους οποίους ο αθλητισμός είναι κομμάτι της καθημερινής ζωής τους και πρέπει να δράσουμε πριν να καταστραφεί η ακαιρεότητα του του σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μποσκούρτ. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω λόγω της σημασίας ε, που παίζει ο αθλητισμός για τους πολίτες της Ευρώπης και της χώρας μου. Ο κύριος Νιούτον Τάν έχει ζητήσει το λόγο. Μπιλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, ε, απευθύνομαι στον πολύ ενδιαφέροντα ομιλητή της Σάντοκ αλλά αναρωτιέμαι εάν ε, οι δύο υπερδυνάμες οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα φοβούνται τόσο πολύ ότι θα πληγεί η ηγεμονία τους ώστε δεν συνεργάζονται. κάνω λάθος, ελπίζω να κάνω λάθος. Επίσης η συγγήτρια που μόλις ε, μας παρουσίασε το θέμα της ε, φαίνεται ότι εννοεί ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε από τον αθλητισμό δηλαδή στις μεγάλες ποδοσφαιρικές ε, ομάδες ε, κανένα θέμα ακόμη και λεπτομέρειες τι ώρα, σε πόση ώρα θα πετάξουν την ε, μπάλα ή θα βγει φάουλ και για να έχει κανείς ένα επιπλέον κέρδος μπορεί να βγάλει την μπάλα φάουλ μετά από 2-3 λεπτά. Ε, αυτό όμω που είναι ανησυχητικό είναι η φλιαρία στο διαδίκτυο. Ε, όταν ε, δείτε ότι υπάρχει μια τέτοια κίνηση ανάβει το διαδίκτυο όπως ε, βλέπαμε πριν από την 11η ε, Σεπτεμβρίου τους διπλούς πύργους υπάρχει τρόπος δηλαδή έτσι να εντοπίσει κανείς τα ανησυχητικά φαινόμενα αυτή είναι η ερώτησή μου ο κύριος Μίτσελ Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε που καθυστέρησα γιατί παρουσίαζα σε μια άλλη επιτροπή μία έκθεση αλλά παρακολουθώ το θέμα ε, σας και ε, ξέρω ότι εάν υπάρχει ε, κάποια, κάποιο παράπτωμα ναρκωτικά κτλ μπορεί να χάσετε ένα βραβείο όπως έγινε παραδείγματος χάρη με έναν σημαντικό αθλητής στις Ηνωμένες Πολιτείες προσφάτως. Αυτό όμως πώς θα το αξιολογούσατε στη συγκεκριμένη περίπτωση αν κάποιος κάνει ζαβολιές ε, και πιστεύετε ότι το άτομο αυτό θα πλήξει την ομάδα του δηλαδή θα χάσει την ε, θα κυριωθεί ο αγώνας για την ομάδα ε, υπάρχει δηλαδή κάποιος πιο θετικός τρόπος να μπορέσουμε να πατάξουμε αυτές τις ε, κινήσεις. Αν δεν υπάρχουν ε, άλλα ερωτήματα, έλεγα λοιπόν ότι εάν δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα, αν δεν δώσω τον ε, λόγο στον εισηγητή θα ήθελα να το ρωτήσω ποια είναι η θέση των κρατών μελών. και να ρωτήσω κυρίως ποια είναι η δική σας άποψη όταν ε, βλέπουμε τέτοιες ε, καταστάσεις ε, να μην ξεχνάμε ότι οι γενικοί αθλητές κυρίως όταν μιλάμε για πρωτοθλητές λαμβάνουν πάρα πολύ ψηλές αμοιβέ και έχουν συμβόλαια πάρα πολύ σημαντικά, κάνουν διαφημίσεις έτσι λοιπόν ε, συνεχίζουν να είναι σημεία αναφορά στο συλλογικό φαντασιακό, θεωρούνται μύθοι. Έτσι λοιπόν ε, με ποιο τρόπο μπορούμε να παρέμβουμε για να αποφύγουμε όχι μόνο να συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις στον αθλητισμό, γιατί πολλές φορές ε, θεωρείται ότι δεν ε, έχουν και σημασία αυτά τα φαινόμενα. Δυστυχώ όμως με ποιο τρόπο μπορούμε να παρέμβουμε για να κάνουμε κατανοητό ε, στα κρατημέλη ότι αυτές οι καταστάσει είναι πάρα πολύ σημαντικέ και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και στη χώρα μου υπήρξε ένα τρομακτικό, απίστευτο σκάνδαλο και τα μέσα μαζική ενημέρωση αναφέρονται μόνο στι σελίδε του αθλητισμού για το θέμα αυτό, ενώ μιλάμε για διαφθορά, για εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε για έγκλημα. Έτσι λοιπόν, κατά τη δική σα άποψη, πώ είναι δυνατόν να παρέμβει κανεί. Και δεν λέω να ευαισθητοποιήσουμε τα κρατημέλη γιατί νομίζω ότι είναι παράδοξο να πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο όρο. Αλλά πώς ε, μπορούμε να απευθυνθούμε στα κράτη-μέλη ε, έτσι ώστε να μην περνάνε σε δεύτερο πλάνο τέτοια ζητήματα σχεδόν απαρατήρητα. Έτσι λοιπόν θα δώσω το λόγο στον κύριο Φυσικό και κατόπιν στην ΕΜΗΝΕ για να απαντήσουν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και ξεκινώ με το επίπεδο διεθνής συνεργασίας στην περίπτωση πολυμερών συνεργασιών. Παραδείγματος χάρη το αναφέρθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που ε, ε, αν χρησιμοποιεί αυτό τον τρόπο στη διεθνή συνεργασία και αν μπορεί να υπάρξουν απελάσεις ε, ή κατασχέσεις βάσει αυτών των μέσων ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων ή στην ε, συνθήκη από διάφορα μέρη του κόσμου. Πολλά έχουν γίνει για να ενταθεί ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων αλλά αυτό είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα και θα αξιολογηθεί τα επόμενα χρόνια βάσει ενός μηχανισμού που θα δημιουργηθεί για να αναθεωρηθεί ε, η συνθήκη και τα πρωτόκολλά της μεταξύ των συμμετοχόντων. Είναι δηλαδή κάτι στο οποίο αναφέρεται εις την συνθήκη του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς. Βεβαίως οι, οι ύποπτες κινήσεις στο διαδίκτυο μπορεί να υποδηλούν ότι κάτι δεν πάει καλά και ε, χρειάζεται όμως ε, ειδικότητα για να μπορεί κανείς να εντοπίσει και να απομονάσει ορισμένες ενδείξεις υπόπτων ε, κινήσεων για παράνομη, παράνομα στοιχήματα παραδείγματος χάρη και είναι ένα θέμα που που πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά και να ε, εντείνουμε την προσοχή μας και αυτό θέτει και το θέμα της αυξήσεως των πόρων και του προσωπικού για να υπάρξουν ειδικές γνώσεις για την ε, ψηφιακή ε, κίνηση σε, ορισμένες, ορισμένα θέματα. Ε, δύο είναι τα θέματα που είναι ενδιαφέροντα. Ε, τα ε, θετικά και βοηθητικά, οι βοηθητικές κινήσεις και η απομόνωση των στημένων παιχνιδιών σε συνδυασμό με την ποινικοποίηση και τον εντοπισμό, την την έρευνα και την δίωξη ορισμένων εγκλημάτων. Δεν είναι μόνο θέμα συνειδητοποίησης, αλλά είναι και θέμα πολιτικής θελήσεως και αποφασιστικότητας. Αν υπάρχει αυτή η αποφασιστικότητα και αιμονή, τότε θα μπορούσε να καταρτιστεί κάτι τέτοιο για να αποδειχτεί η αποτελεσματικότητα και των προληπτικών πολιτικών και ε, των αντιδράσεων της δικαιοσύνης στα στημένα παιχνίδια σημαίνους αγώνες δηλαδή. Ε, θα ήθελα επίσης, αν μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, να σχολιάσω τις ε, συστάσεις οι οποίες ε, πρότεινε προηγουμένως ε, η κυρία Μπόσκουρτ. Νομίζω ότι ο κατάλογος αυτός αναφέρεται σε πολύ ε, χρήσιμα στοιχεία, καλύπτει πάρα πολλούς εμπλεκομένους και ενδιαφερομένους, να μην υπάρχει καμία ανοχή για τη διαφθορά παραδείγματος χάρη η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με τα στημένα παιχνίδια και με τα ε, στοιχήματα και είναι όμως θέμα μεταξύ των ε, αρχών ε, διατήρησης ε, εφαρμογής της τάξης νομικών αρχών και του ιδιωτικού τομέα και επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί η νομοθεσία των κρατών κατά τρόπον ώστε να υπάρξει μια πιο στενή συνεργασία. Εφόσον λοιπόν είναι σημαντικό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα όλων των μέτρων που αναφέρονται εις την ποινικοποίηση θα χρειαστεί μία συνολική αντιμετώπιση και προσέγγιση από όλους τους ε, ενδιαφερομένους για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Ευχαριστώ, η Εμινέ Μποσκούρτ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις καλές ερωτήσεις τους και ναι, για την πρώτη ερώτηση ε, μπορείτε να στοιχηματίσετε σε οτιδήποτε. Αν το εξετάσετε, τα στοιχήματα αυτά καθεαυτά δεν είναι αυτά που δημιουργούν το πρόβλημα στοιχήματα ένας τρόπος ξεπλήματος ε, χρημάτων και το βασικό είναι τα στημένα παιχνίδια, ο εκφοβισμός, η δωροδοκία των παικτών και ούτω καθεξής. Βεβαίως μπορείτε να κάνετε πολλά σε συνεργασία με τις εταιρείε που διαχειρίζονται τα στοιχήματα διότι αυτές θέλουν να διατηρήσουν το λόγο υπάρξεό τους Οπότε ε, είναι πολύ καλό ότι τώρα ε, έχουν εμπλακεί στην παρακολούθηση με ε, υπομνήματα συνεργασίας γιατί όπως είπα στην εισαγωγή μου θα βοηθούσε να υπάρχει και ένας κώδικας συμπεριφοράς σχετικά με τα στοιχήματα. Όσον αφορά δε τη μηδενική ανεκτικότητα κατά της διαφθοράς, ε, ε, είτε εντός είτε εκτός οργανώσεων, Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτοί που εμπλέκονται στις ε, οργανώσεις να μην, ε, είναι, ε, να, μην μπορούν να δοκιθούν και χρειάζεται μία νέα προσέγγιση και έρχομαι έτσι στη δεύτερη ερώτηση τι θα γίνει αν υπάρξουν ποινές πρέπει να τιμωρούνται και οι όμιλοι, οι ομάδες, βεβαίως. Καμιά φορά Πριν από μερικούς μήνες, παραδείγματος χάρη, η, παρουσιάστηκε η μαύρη βίβλος για το ποδόσφαιρο των ανατολικών χωρών, όπου από πλευράς στημένων παιχνιδιών και διαφθοράς και διαρροών υπάρχουν πολλά προβλήματα, οπότε για να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να τους τιμωρήσουμε και αυτούς. Όταν όμως εμπλέκονται μόνο παίκτες ή διαιτητές, τότε μόνο αυτά τα άτομα θα έπρεπε να εμπλακούν και αυτό είναι λογικό. Αλλά αυτό μπορούν να κάνουν οι ομάδες είναι να αυξήσουν την πρόληψη ιδίω για τους νέους παίκτες να τους ε, εκπαιδεύσουν να τους ε, συνειδητοποιήσουν εναντίον των στημένων παιχνιδιών γιατί σχετικά με το τελευταίο ερώτημα της Προέδρου Δεν είναι οι παίκτες ε, με τους τεράστιους μισθούς οι οποίοι είναι ευάλωτοι στα ε, στημένα παιχνίδια αλλά από όταν, ε, από ό,τι φάνηκε από τη μαύρη βίβλο του ποδοσφαίρου ανατολικών χωρών είναι αυτοί που έχουν ε, μικρούς μισθούς, δυσκολίες ε, και δεν τα βγάζουν πέρα ή οποίοι στείνουν τα παιχνίδια και ε, εμείς βλέπουμε μόνο τους δημοφιλείς παίκτες αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Πέρυσι όταν έγινε το Συμβούλιο των Υπουργών Αθλητισμών το Νοέμβριο αυτό που, ήρθε, που δημοσιεύθηκε ως αποτέλεσμα του Συμβουλίου Υπουργών Αθλητισμού δεν ήταν πολύ συγκεκριμένο Οπότε ε, θα πρέπει να υπάρξει μία πρόταση για το επίσημο Συμβούλιο Υπουργών Αθλητισμού και να προβούν ε, σε ένα ορισμό των στημένων παιχνιδιών ε, και των προβλημάτων στον αθλητισμό κατά τρόπον ώστε σε συνδυασμό με την τις αστυνομικές αρχές να μπορέσει κανείς να επιτύχει διότι δεν είναι μόνο ότι καταστρέφουν το ποδόσφαιρο αλλά είναι σοβαρή, ε, σοβαρές κινήσεις του υποκόσμου, της μαφίας και γι' αυτό και στα κράτη-μέλη μας θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να κινηθούν διότι μέχρι στιγμής πιστεύω ότι δεν, είναι, δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί όλες οι χώρες για να κάνουν κάτι για να πατάξουν το φαινόμενο αυτό και έχει φτάσει η ώρα να το λύσουμε σαν θέμα. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι σε αυτά που ανέφερα πριν και να απαντήσω στην ερώτηση στα είδη προδραστικών μέτρων. Δηλαδή όπως ε, η καθαίρεση κάποιων αθλητών ε, ή ε, η ακύρωση κάποιων αθλητικών εκδηλώσεων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει, αλλά αυτό εξαρτάται από το βαθμό της υποψίας που υπάρχει για το αν αυτή η αθλητική εκδήλωση, αυτό το αθλητικό γεγονός θεωρείτε ότι, ότι θα μπορούσε να είναι στημένο. Και ο βαθμός ε, της υποψίας είναι νομοθετικό ζήτημα, αν υπάρχει ασφάλεια δικαίου ότι ε, δηλαδή αποφεύγεται κάθε είδος ε, αυτεριστής, τότε αυτά τα προδραστικά μέτρα θα μπορούσε να είναι κάποιες επιλογές Και θα μπορούσαμε να έχουμε λοιπόν τέτοια προληπτικά μέτρα κατά του στισίματος αγώνων. Αλλά θέλω να θέσω ένα θέμα. Γιατί μιλήσαμε για την ανάγκη εναρμόνιση ε, των εθνικών ε, προσεγγίσεων ως προς την ποινικοποίηση και την ε, δυνατότητα ενός νέου μέσου, μιας νέας οδηγίας, όπου πιθανόν να περιλαμβάνεται και ένας ορισμός. Και ουσιαστικά εγώ μοιράστηκα την εμπειρία μου μαζί σας από ένα διαφορετικό πολυμερές πλαίσιο από τον ΟΗΕ. Και φυσικά αυτό σχετίζεται και με αυτό που συζητήσαμε για ένα πιθανό ορισμό για το έγκλημα στον κυβερνό χώρο. Πριν να ξεκινήσουμε να συζητάμε τα, θέματα, τα άλλα θέματα όταν ε, επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά ε, στους ορισμούς των εγκλημάτων αυτό θα μπορούσε να είναι αντιπαραγωγικό ενίοτε γιατί θυμάμαι ότι στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων και τη ε, σύμβαση του Παλέρμο για το Διεθνές Οργανωμένο και για τη σύμβαση κατά τη διαφθοράς τα θέματα του ορισμού των εγκλημάτων τέθηκαν και η τελική λίστα να μην συμπεριληφθούν ορισμοί των αδικημάτων, αλλά ή να έχουμε ορισμό των δραστών ή να έχουμε μία πιο περιγραφική προσέγγιση ποινικοποιώντα ένα σύνολο περιπτώσεων. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να δούμε αν μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. καθώς ε, οι συζητήσεις ε, για την ορολογία μπορεί να επιφέρουν πρόσθετες δυσκολίες και πιθανές συγκρούσεις. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, εγώ φοβάμαι ότι οι πτυχές αυτές θα μπορούσαν ε, να χρησιμεύσουν ε, στο να μην εκπαιδευτούμε στο πραγματικό πρόβλημα. Ένα δίκημα είναι ένα δίκημα και κατά την άποψή μου για να αντιμετωπίσουμε τη μαφία και τον οργανωμένο έγκλημα θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να ορίσουμε το αδίκημα αυτό χωρίς να αφήνουμε σε κανένα τη δυνατότητα να το ερμηνεύσει. Και το επαναλαμβάνω, οι εγκληματίες ξέρουν πολύ καλά τι ξέρουν και τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Για αυτούς είναι σαφές, ενώ εμείς πολλές φορές χάνουμε πολύ χρόνο στο να καταλάβουμε πώς θα κινηθούμε και πολύ συχνά από έξω οι πολίτες μπορεί να έχουν την εντύπωση ότι οι νομοθέτες περιστρέφονται γύρω-γύρω από το θέμα και δεν θέλουν ε, τελικά να αναλάβουν δράση. Εγώ θεωρώ ότι ένα δίκημα παραμένει ένα δίκημα και το ξαναλέω γιατί εσύ στις απαντήσεις σου έμεινε είπες ότι συχνά ε, αυτοί που πέφτουν στα δίχτυα της διαφθοράς ε, και των παρόμοιων στιγμάτων και αυτά είναι αυτοί που δεν έχουν υψηλούς μισθούς, παίκτες που δεν έχουν υψηλούς μισθούς. Εγώ θυμάμαι ότι άκουσα ένα πάρα πολύ διάσημο παίκτη στη χώρα μου ο οποίος είπε ότι αισθανόταν ότι μπορεί ελεύθερα να στοιχηματίσει ένα εκατομμύριο ευρώ. Σαν να ήταν ε, απόλυτα μια απόλυτα κανονική πράξη και αυτό δεν ε, διακινδυνεύει μόνο να γίνει πρακτική αλλά μια σχεδόν κανονική συμπεριφορά, μια συμπεριφορά που θα επιτρέπεται. Ενώ εγώ αντίθετα θεωρώ ότι επί αυτών των πτυχών θα πρέπει να ε, μην υπάρχουν αμφιβολίες ε, για το ποιος πρέπει να είναι ή δεν πρέπει να είναι ο ορισμός του αδικήματος. Θα πρέπει να υπάρχει αδιαλαξία από αυτού και νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσουν άλλο χρόνο τα κράτη-μέλη, γιατί διακινδυνεύουμε ε, εδώ να αφήσουμε να εξαπλωθεί το οργανωμένο έγκλημα στο συγκεκριμένο τομέα. Ευχαριστώ. Του ε, προσκεκλημένου μα, Αν ε, δεν θέλει κάποιο άλλο το λόγο για να προσθέσει κάτι, μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ αυτή τη συνεδρίαση. Και θέλω να υπενθυμίσω στους αξιότιμους κύριους βουλευτέ ότι αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε στις 9 με την ακρόαση του Γενικού Διευθυντή Εσωτερικών Υποθέσεων, τον κύριο Μασερβίση. Έτσι λοιπόν, ε, σα παρακαλώ να έρθετε εδώ εγκαίρως. Θα ξεκινήσουμε στι 9. Καλό σα βράδυ.